Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζου ολοκλήρωσαν πολύ πρόσφατα το πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την νέα εκδοχή της Συμφωνίας Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης η μονογραφή της ε, συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί και θα σας ε, θα υποβληθεί ως ανώπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να εγκρίνουμε τη σύναψη αυτής της ε, αναθεωρημένης συμφωνίας. Έχουμε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα αυτό και άλλωστε καθ' όλη τη διάρκεια του 2012 κάναμε σχετικές συστάσεις και θα αγγίψουμε και στη συμφωνία αυτή σύντομα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη, αλλιώ να περάσουμε στο θέμα τη Μολδαβία. να αλλάξουμε τη σειρά στο 4 και στο 5 αν θέλετε και να κοιτάξουμε πρώτα το θέμα της επικύρωσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίρρηση για να αποφασιστεί μετά το σχέδιο ψηφίσματος με τις ε, τροπολογίες. Έχει για τους ηγητής μήπως παρατηρήσεις να κάνει. Mr. Chairman, colleagues, ladies and gentlemen, indeed, uh, Πρόεδρε, συνάδελφοι, ζητώ την υποστήριξή σας και τη συμφωνία σας σε ό,τι αφορά το σχέδιο αποφάσεων του συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπηρεσίας Ατομικής Ενεργείας και των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ε, Μολδαβία. Νομίζω ότι είμαστε υπέρ τη συμφωνία αυτή και ζητώ την υποστήριξή so, Να περάσουμε όμως τώρα στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Εδώ θα ψηφίσουμε μόνο ναι, όχι οι αποχέ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ηλεκτρονικά λοιπόν. Έναξη ψηφοφορίας. Die Abstimmung ist geschlossen. Der Assoziierungsvertrag η συμφωνία σύνδεσης με την Μολδαβία εγκρίνεται με ψήφους 44 υπέρ, 3 κατά, 0 εποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. και να εκφράσουμε την ελπίδα για μια καλή συνεργασία στα πλαίσια με συμφωνία σύνδεση με τη Δημοκρατία της Μολδαβία. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι υπεύθυνο γι' αυτό ο συνάδελφο Πλέγκοβιτ. Α, συγγνώμη, κύριε Σκούζο. Συνεχίζουμε με την παράγραφο 1 της έκθεσης. Ψηφίζουμε την παράγραφο 1 παρακαλώ. Συμβαστική τροπολογία 2. Συγγνώμη, ήταν η παρθενική μου ψηφοφορία. Διανατάσσεω ισχυρό, υπέρ παρακαλώ, κατά. Εγκρίνεται. 25 καταπίπτει. 26 το ίδιο. 27 το ίδιο. Και 28 καταπίπτει. 29, 30, 32 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την 31 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 33. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ? Κατά. Καταπίπτει. Ε, όχι, μάλλον απορρίπτει. 34 για την παράγραφο 3. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται, μάλλον. Προφορική τροπολογία. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 35. Δεκάει, Δεκάει. Check, Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το τμήμα 2 της προφορικής τροπολογίας. Παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. «26 υπέρ, 29 κατά». Απορρίπτεται. Η 35 καταπίπτει, το ίδιο και η 65. Συμβασική τροπολογία 3 τώρα. Διανατάσω τη χειρός. Παρακαλώ ποιος είναι υπέρ για τη συμβαστική τροπολογία 3. Εγκρίνεται. Επανάληψη της ψηφοφορίας. Σας ζητώ συγγνώμη και πάλι γιατί είμαι καινούριο σε αυτά. Για τη συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απόχες. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 3. Καταπίπτουν 36, 37, 38, 39, 45 και περνάμε στην παράγραφο 5 και την, την τροπολογία 40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται μάλλον. 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 47 προς 9. Πρέπει να σηκώνετε τα χέρια για να μπορούμε να κάνουμε την καταμέτρηση. 44. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Κατά. Απο, κα, απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Τροπολογία 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Καταρρίπτεται. Α, προτιμάτε ηλεκτρονικό έλεγχο. Εντάξει, ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται η τροπολογία 47. Τροπολογία 48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 49 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 49 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 49. 51 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Για την παράγραφο 4, συμβαστική τροπολογία 4, ε, παράγραφος 10, συγγνώμη, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 53, 54, 55, 56 και 57. Θα ψηφίσουμε την 58. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται καταπίπτουν οι 61, 62, 63, 64 και ψηφίζουμε την 66. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι 50, 67 και 68 καταπίπτουν. 69 ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 70 κατά τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα της 70 71 ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 72 υπέρ κατά απορρίπτεται η 72 απορρίπθηκε και ζήτησε το λόγο ο εισηγητής Αυστρεβίτσιος. Πρόεδρε, να στηρίξω την τροπολογία Πρέντα Μακοβέη. Να σας παρακαλέσω να ψηφίσετε υπέρ. Η συμβαστική να εγκριθεί. Για την τροπολογία 73, λέει ο συγκητής, Είμαι υπέρ της τροπολογίας Πρέντα και Μακοβέη, αριθμόν 73. Ψηφίζουμε λοιπόν την 73. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ονομαστική ψηφοφορία λέει ο πρόεδρος. Ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος διορθώνει. Ποιος ψηφίζουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Faltan Ramos. Continuamos. <clears throat> Εγκρίνεται. 74. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 76. Α, συγγνώμη, καταπίπτει λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την 80. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 80. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 81. ένα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 7. Καταπίπτουν οι τροπολογίες 82 μέχρι 89. 90 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 97. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 98. Πρώτο τμήμα. Ακαλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία 8. Ε, 2 υπέρ, κατά. Τμήμα 2 τμήμα 2 της τροπολογίας 98. Επανάληψη ψηφοφορίας. Ποιος είναι υπέρ του τμήματος 2 της τροπολογίας 98. Κατά. Απορρίπτεται. 99. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ κατά απορρίπτεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 7 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 9 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στη 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την προηγούμενη, για την τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. La 15 la habíamos votado, pasamos a Τη 15 την ψηφίσαμε, περνάμε στη 16. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 16. 16. Ελεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι τροπολογίες 18 έως 22. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 22. Κατά. Απορρίπτεται. 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται. Περνάμε στην 24. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Θεωρώντας. 1. Τροπολογία 1. Στο θεωρώντας 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Για την πρώτη παράγραφο, ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 1 είναι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 είναι κατά πίπτη καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία 8. Τροπολογία 3 είναι τα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Είναι τα 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Είναι τα 5. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Είναι τα 6. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την πέμπτη τροπολογία της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τροπολογία 5 της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου. Τέσσερις δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 είναι τα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 7 της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία 7. Ηλεκτρονικός έλεγχος τώρα για την προηγούμενη τροπολογία, την 6 της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6, άρχεται η ψηφοφορία. Πάσα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 τώρα της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά της 8. Εγκρίνεται. ΙΝΤΑ 9. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. ΙΝΤΑ 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πρέπει τώρα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Απρόβαδο. Εγκρίνεται. Hemos acabado con los votos. Discúlpenme, pero mi Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Σα ζητώ συγγνώμη που σα είπα, ήταν η παρθενική μου ψηφοφορία. Σίγουρα τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερο. Empezamos en un minuto, dos minutos. Σε ένα-δύο λεπτά συνεχίζουμε. Σε ένα λεπτό θα συνεχίσουμε. Έχουμε την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γεωργίας στη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Τέα Τσουλουκιάνη, που είναι Υπουργός Δικαιοσύνης της Γεωργίας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται να κάνουμε συζήτηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γεωργίας. Κύριε Υπουργέ, είχαμε ανταλλαγή απόψεων και πριν από ένα χρόνο περίπου και τότε μας ενημερώσατε για το πρόγραμμα της κυβέρνησης ε, της Γεωργίας για, την, ε, για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ετοιμορρησίας. Τον Ιούνιο συνυπογράψαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Συμφωνία σύνδεση ε, που κυρώθηκε από τη Βουλή σα και θα συζητηθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, έγινε εναρμόνιση των θεωρήσεων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε και την έκθεση του Ιουλίου του 2014 του κ. Τόμα Χάμεμπαρ που είναι ο ειδικό συζητητή Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη στη Γεωργία. Και η έκθεση αναγνωρίζει την πρόοδο τη Γεωργία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προβαίνει και σε πολλέ συστάσει. Είμαστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση της Γεωργίας θα τις λάβει υπόψη και με κυρίαρχο τρόπο θα λάβει μια θέση. Βέβαια είδαμε ότι πρόσφατα κατηγορήθηκαν ε, πρώην αξιωματούχοι και ο πρώην πρόεδρος Σακασβίλη. Βέβαια, εμεί έχουμε εμπιστοσύνη ότι η Γεωργία και η δικαιοσύνη της, η δικαστική τη εξουσία θα αποφασίσουν με επιμέλεια για να αποφασίσουν αν αυτοί οι αξιωματούχοι και ο πρώην πρόεδρος Σακασβίλη είναι αθώοι ή ένοχοι. Οι μεταρρυθμίσει στη Γεωργία τη χάνουν ε, μεγάλης προσοχής και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να σας δώσουμε αμέριστη υποστήριξη είναι να έχουμε εμπιστοσύνη αμοιβαία. Θα σας δώσω το λόγο για ένα δεκάλεπτο για να μας παρουσιάσετε το δικαστικό σύστημα της πατρίδας σας, της Γεωργίας. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, είναι τιμή μου που μπορώ να λάβω το λόγο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα. Είναι και μια μεγάλη ευκαιρία επίσης να δούμε μαζί που έχει φτάσει ως προς τις ευρωπαϊκές τη προσδοκίες η Γεωργία. Θα θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου είχα έρθει και πάλι εδώ εξηγώντα πώ θα εκτελέσει τις μεταρρυθμίσεις που αναμένονται από εμά η Γεωργία. Και εξηγώντα ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να είναι τελεσίδικος και για όλε τι επόμενε κυβερνήσει. Γι' αυτό λοιπόν ένα χρόνο μετά αποφάσισα, επειδή υπάρχουν εξελίξεις, να ξανάρθω και σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Είναι ενθαρρυντικό να συζητούμε με όλες και όλους εσάς τις μεταρρυθμίσεις μας. Πρόεδρε, ως προς την υλοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης και του προγράμματος απελευθέρωσης αλλά και περαιτέρω. Είναι σημαντικότατα εργαλεία που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές αρχές να ισχύσουν στο νομικό και δικαστικό πλαίσιο της Γεωργίας. Είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος ε, η συνεργασία αυτή και να εξηγήσω πώς. Η Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία διευρύνει τις ρυθμιστικές ε, ε, δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και με την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής η απόσταση που μας χωρίζει μικραίνει. Οι δημοκρατικοί θεσμοί θα πρέπει να εδραιώσουν περαιτέρω το δημοκρατικό σύστημα στη Γεωργία για να γίνει μια χώρα σταθερότερη και ένα παράδειγμα δημοκρατικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή με πολλά προβλήματα αυτό το διάστημα από την Ανατολική Ουκρανία στο Ιράκ και τη Συρία. Οι νομικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις πιστεύω ότι ενισχύουν και ενδυναμώνουν τη δημοκρατική σταθερότητα και ασφάλεια στη Γεωργία. Και με τον ίδιο τρόπο οι κανόνες που βασίζονται στην ε, διεθνή τάξη και την διεθνή ασφάλεια. Η επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος είναι σημαντική και για μας για εσωτερικούς λόγους. Βέβαια υπάρχουν αμφιβολίες από τους ευρωσκεπτικιστές. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένη στη διεθνή δημοκρατική σταθερότητα και το διεθνές ε, δίκαιο προσφέρει τις ε, πολλές νέες δυνατότητες στη χώρα. Ο εξοπλισμός της χώρας ε, της Γεωργίας δεν είναι πλέον κάτι το αντιστρέψιμο και πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο των υποσχέσεων ευθυγραμμιζόμενοι με τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και την καλή διακυβέρνηση, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαστικό σύστημα, χωρί να παραμένει κανένα ε, ενδιασμό καμία αμφιβολία. Σε αυτό το πλαίσιο η υπογραφή τη Συμφωνία Σύνδεση ήταν μεγάλη σημασία, ήταν ένα θετικό βήμα προόδου για να ε, συνεχίσει αμετάκλητη αυτή η πορεία προς την πολιτική μας σύνδεση και την οικονομική ε, ένωση με την Γεωργία ώστε να γίνει ένα μη επίσημο, αλλά ε, επίσης τρόπον την συνεργαζόμενο κράτος μέλος η Γεωργία. Η προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 επέτρεψε σε ένα μεγάλο μέρο των αρχών, προτύπων και ρυθμίσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματωθούν στο δικό μα νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική η διαδικασία τη υλοποίηση των ευρύτατων μεταρρυθμίσεων που αναμένονται. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι από την πλευρά μα, η κύρωση τη συμφωνία, δεν ήταν ο απότατο ε, στόχο, ούτε αυτό ο σκοπό. Ήταν ένα πραγματικό μαραθώνιο που πρέπει να μα οδηγήσει στην ευρύθμη λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος των δημοκρατικών θεσμών στη Γεωργία. Η πραγματική ε, υλοποίηση της συμφωνίας ε, πρέπει να γίνει με κοινή ανάληψη ευθύνη και είναι σημαντική για την εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων από την πλευρά μας. Έχουμε προβλέψει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο. Ιδιαίτερο η κυβέρνηση έχει αναβαθμίσει του εσωτερικού μηχανισμού συντονισμού. Επίση έχει επεξεργαστεί ένα εθνικό πρόγραμμα δράση για την συμφωνία σύνδεση και την υλοποίησή τη και ένα τριετέ πρόγραμμα δράση για την ε, συμφωνία αυτή της απελευθέρωσης των ε, εμπορικών συναλλαγών. Είναι μια ε, απαιτητική διαδικασία βεβαίω αυτή και θα εξαρτηθούν πολλά και από τη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κατών μελών να στηρίξουν τις προσπάθειές μας και να προσφέρουν τεχνική αρρωγή βάσει των αρχών της διαφυροποίησης και του more for more, περισσότερα για περισσότερα. Ξεκίνησα τον, ε, την ομιλία μου μιλώντας για τα εγχειρήματά μας και την προσπάθεια να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας. Οι πρώτες φάσει της, του προγράμματος δράσης απελευθέρωσης έχει ξεκινήσει. Την περασμένη χρονιά είχα την ευκαιρία να σας ε, μιλήσω και πάλι και να σας πω ότι θα υλοποιήσουμε εγκαίρως το πρόγραμμα δράσης. Σήμερα μπορώ με καμάρι να σας πω ότι η Γεωργία έχει εκπληρώσει τις βασικούς όρους τη υλοποίηση του προγράμματο δράση και ήδη έχει περάσει στη δεύτερη φάση και τι προτεραιότητέ τη. Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε πλήρω το σύστημα με την συγκριτική αξιολόγηση, με αυτά που προκύπτουν από την Σύνοδο τη Ρήγα. Ε, από τη Σύνοδο της Ρήγας και να περάσουμε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην πλήρη υλοποίηση, στη δεύτερη φάση του προγράμματος απελευθέρωσης. Επίση, θα πρέπει να υπάρξει και απελευθέρωση του καθεστώτο θεωρήσεων. Αυτή η απελευθέρωση έχει πολύ σημαντική πολιτική διάσταση και για μα. Ε, το ξέρετε αυτό. Θα γίνουν τα γεωργιανά διαβατήρια πιο ελκυστικά βεβαίω και από κατεχόμενα εδάφη. Και όπω έχει σημειωθεί, πρέπει να μοιραζόμαστε τι ίδιε αρχέ και αξίε. Ε, τη δημοκρατία, την καλή διακυβέρνηση, την διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό του. Όλα αυτά είναι ε, ύψης της σημασίας για να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Γι' αυτό ήθελα να αναφέρω τα κύρια επιτεύγματα της γεωργίας το πρόσφατο διάστημα. Πρώτα απ' όλα για τι εκλογέ. Το βασικό επίτευγμα για τις πρόσφατες εκλογέ, κοινοβουλευτικέ το 2012, προεδρικέ το 2013 και δημοτικές το 2014. Εδώ καταφέραμε να αποσυνδέσουμε το, τη λειτουργία των βασικών ε, κομμάτων από το κράτος. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον συγχώνευση κρατών, του κράτους με το κυβερνών κόμμα. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και η Ομάδα Δράσης για τις Ελεύθερες Εκλογές επιτρέπουν με τη λειτουργία τους να μην υπάρχει ε, ανεπιθύμητη επίδραση των πολιτικών ευθυνόντων στην προκλητική εκστρατεία και την εκλογική διαδικασία. Επίσης, τις ημέρες των εκλογών καταφέραμε να έχουμε ελεύθερες ε, διαδικασίες, ελεύθερη ψηφοφορία των πολιτών. Και έχει γίνει πλέον η εκλογική διαδικασία μια δημοκρατικότατη και πάγια ε, διαδικασία. Το Συμβουλίο της Ευρώπης μάλιστα πρόσφατα δημοσίευσε μια δήλωση αποτιμώντας τις εκλογές του 2014 στη Γεωργία και είναι πολύ θετική η αξιολόγηση αυτή. Τώρα τομεακέ μεταρρυθμίσεις. Μέρος των πρωταρχικών στόχων να έχουμε ένα εύρυθμο δημοκρατικό σύστημα στη Γεωργία ήταν η υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας ε, του κράτους δικαίου, της ε, ε, επιβολής του κράτους δικαίου και της εδώ συμπεριλαμβανόταν το ειρήνη στη Γεωργία, ε, κυρίως ε, στις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν. Ήταν προτεραιότητα η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και θα θυμάστε και πέρσι σας τα εξέθεσα και σας τα ανέφερα. Η πρώτη φάση ήταν η αποπολιτικοποίηση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γεωργίας, ώστε οι πολιτικοί και οι παρήσακτοι να φύγουν από το δικαστικό σύστημα, να απελευθερωθεί ο δικαστικός κλάδος από εξωτερική πίεση ή επιρροή. Το δεύτερο κύμα των μεταρρυθμίσεων αφορούσε ένα ελευθερότερο και ανεξάρτητο σύστημα εκλογής των δικαστών, και η τρίτη φάση αφορά την ε, εσωτερική ανεξαρτησία των δικαστών και την ανάθεση εξουσιών μέσω της δικαστικής τους λειτουργίας, του δικαστικού τους λειτουργήματος. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την τοποθέτησή τη για τι τρει φάσει των μεταρρυθμίσεών μα και η αξιολόγηση τη ήταν και πάλι θετικότατη. Πρέπει όμω τώρα να ενσωματωθούν οι συστάσει τη Επιτροπή τη Βενετία σε διάφορα μέρη της νομοθεσίας μας και να να προχωρήσουμε στην τρίτη φάση μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη ήταν μια άλλη προτεραιότητα. Η νέα νομική υπηρεσία που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, τη λογοδοσία και την διαφάνεια της, ε, του όλου συστήματος και παρέχει κοινωνικές εγγυήσεις για του κοινωνικού εταίρου. Είναι διαφορετικό από το Υπουργείο των ε, Ποινών και των ε, Φυλακών οι υπηρεσίες ε, ανήκουν πλέον σε έναν εξάρτητο φορέα που είναι ε, υπεύθυνο να λογοδοτεί ενώπιον του Κοινοβουλίου. Η θεσμική ανεξαρτησία των εισαγγελικών αρχών και η αμεροληψία τους, η απελευθέρωση από την πολιτική επιρροή ήταν πολύ σημαντική προτεραιότητα. Το πρώτο βήμα έγινε τον Μάιο του 2013 και οι πλήρες εισαγγελικές ε, αρμοδιότητες ανατέθηκαν στον επικεφαλής ε, εισαγγελέα της ε, χώρας. Οπότε εγώ η ίδια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Υπουργό Δικαιοσύνης δεν μπορώ να παρέμβω καθόλου σε οποιαδήποτε υπόθεση απλώς με τον πρώτο εισαγγελέα της χώρας, το Γενικό Εισαγγελέα της χώρας μπορώ να προβλέψω κατευθυντήριες γραμμές απλώς για την υπηρεσία των, ε, την εισαγγελική υπηρεσία της χώρας με κάποιες βασικές συστάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως. Είχαμε πάντοτε από πολλά χρόνια προβλήματα στις αίθουσες των δικαστηρίων της ίδιας στη Γεωργία. Θυμάμαι όταν εγώ εργαζόμουν ε, σε υποθέσεις γεωργιανών ο ποινικό μα κώδικα δεν εξασφάλιζε την, την αμερόληπτη εκδίκαση των υποθέσεων. Γι' αυτό εγκρίναμε στόχους που εγκρίνουν την ε, εκδίκαση υποθέσεων δια που επηρεάζουν όλων των ειδών της υποθέσεις. Θα θυμάστε ότι στη Γεωργία ποινική μας δικαιοσύνη δεν βασίζεται στην, ε, στην ε, ανακριτική, στο ανακριτικό σκέλος, αλλά με τις τροπολογίες που επιφέραμε, ουσιαστικά μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε να μην είναι η υπεράσπιση λιγότερο δυνατή από την εισαγγελία. Είναι πλέον ισότιμη η εκπροσώπησή τους ε, στην ε, στις δικαστικές αίθουσες. Οι δίκες επίσης με ενόρκους ήταν μια καινοτομία που προβλέφθηκε στο δικαστικό σύστημα στη Γεωργία. Ήταν μια από τις προτεραιότητες της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν είχαμε τέτοιου είδους ε, πείρα, εκτός από το σύντομο διάστημα ανεξαρτησίας της δημοκρατίας της Γεωργίας πριν γίνει η Σοβιετική Δημοκρατία η Γεωργία μεταξύ του 1918 και 1921. Προτού το σύστημα αυτό διευρυνθεί και πριν συμμορφωθεί πλήρως με τα πρότυπα ECA, θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθίες μας. Η μεταρρύθμιση λοιπόν του συστήματος επιτρέπει να μην υπάρχει ένα παζάρεμα από τις εισαγγελικέ αρχές που να εκδικαστεί μια υπόθεση. Ε, αυτό ίσχυε από πολλά χρόνια, από το 2004. Ε, οι δικαστικοί διακανονισμοί λοιπόν οργανώνονται πλέον διαφορετικά και η όλη διαδικασία ε, οργανώνεται ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Έχουμε προβλέψει την έννοια του πρωτοκόλου σήμερα όπου πρέπει να καταγράφονται από τις δικαστικές υπηρεσίες τα πρακτικά των δικαστικών διακανονισμών για να είναι όλα ουδέτερα. Τώρα για τα δικαιώματα των ε, θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες προβλέψαμε από, τη θυμάστε ήταν προτεραιότητα του Υπουργείου μας και από την προηγούμενη ομιλία μου φάνηκε αυτό, προβλέψαμε συγχρονότερα πρότυπα για τα δικαιώματα των θυμάτων, ευρωπαϊκά πρότυπα και σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, αλλά και σε βάση των βέλτιστων πρακτικών που διεθνώς ισχύουν. Ο σχετικός νόμος εγκρίστηκε τον Ιούλιο φέτος, ε, από το Κοινοβούλιο μας βάσει της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2012 για την προστασία των θυμάτων ε, και βάσει των όσων ισχύουν και μέσω της δικαιοδοσίας του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Από το 2011 λοιπόν έχει ξεκινήσει η σχετική προσπάθεια και έχουν αναγνωριστεί οι προσπάθειές μας για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και τη διαφάνεια και τον 2014 εκλεγήκαμε ως μέλος της ε, Διευθυντικής ε, της ε, Επιτροπής Καθοδήγησης του OGP. Αυτό ασχολείται και με τις με την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτά είναι, αυτό είναι το πλαίσιο εντό το οποίο ασχολούμαστε και από το Σεπτέμβριο του 2014 είναι ε, υποχρεωτικό από το νόμο ηλεκτρονικός να αποκαλύπτονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, οι κρατικές δομές μπορούν να λειτουργούν καλύτερα και με, διαφανές, με διαφανή τρόπο, εφαρμόζοντας το σύστημα παροχής πληροφοριών διεθνή πρότυπο. Εδώ θελήσαμε να εξασφαλίσουμε και την ε, ε, προστασία όσων αποκαλύπτουν πληροφορίες εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα με σχετική παρέμβαση του Τμήματος Αστικού Κώδικα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρθηκε από τον ε, Πρόεδρο πριν από λίγο, η πρώτη εθνική στρατηγική και πρόγραμμα δράση τη Γεωργία για το θέμα αυτό εγκρίθηκαν το, από το Κοινοβουλίο τον Απρίλιο του 2013 και τον Ιούλιο του 2013 αντιστοίχω. Έχουμε πλέον μια επταετή στρατηγική για την εθνική στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου υπάρχει μια διαδικασία με συμμετοχή κρατικών φορέων και διεθνών οργανισμών. Η στρατηγική αυτή χαράχτηκε βάσει της ε, των συμπερασμάτων του, Διεθνούς του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του, της Εισαγγελικής Υπηρεσίας και βεβαίως των συστάσεων του Ευρωπαίου Πρέσβη στην ε, παρατηγορία του κ. Τόμας Χάμερμπεργκ. Υπήρξαν και άλλες δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Ε, τον Ιούλιο του 2013 εγκρίθηκε ο σχετικός νόμος για την αντιμετώπιση της μη διακριτικής μεταχείρισης βάσει του φύλου, ε, της ε, εθνοτικής προέλευσης, της ταυτότητας, των σεξουαλικών προτιμήσεων, της υγικής κατάστασης και ούτω καθεξής. Και, στη δημοτική, και, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο προκειμένου να υπάρχει προστασία των δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε μορφή διακριτικής μεταχείρισης βάσει αυτού του νόμου, έμεση ή άμεση ή πολλαπλή, απαγορεύεται. Επίσης για τη στατηγική εξέταση των προσφυγών και των κανόνων που ισχύουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, ήδη την τελευταία πενταετία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα πρότυπα και για να καταλάβετε πόσο έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο Γεωργιανό δικαστικό σύστημα, να, καταλα... να δείτε ότι όταν είχαμε περίπου 200 προσφυγές το πρώτο εξάμεινο το 2010-2011 και 2012 φέτος φτάσαμε μόνο στις 79 αντιστοίχω. και κλείνει το πρώτο εξάμενο μάλλον πέρσι το 2013 είχαμε μόλις 79 και φέτος έχουμε 50 αυτό δείχνει πόσο έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα Από ό,τι καταλαβαίνετε από την παρουσία, παρουσίασή μου, οι αριθμοί δείχνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές στο δικαστικό σύστημα της Γεωργίας, στη δικαιοσύνη γενικότερα, προχωρούν και βελτιώνονται. Δεν θα ακόμα πολλά μπορούν να αλλάξουν, αλλά σήμερα ήθελα να έρθω εγώ να σας ε, εξηγήσω πώ ακολουθήσαμε τι συστάσει σα και τι συμβουλέ σα. Πώ προσπαθούμε να κάνουμε ακόμη ε, ε, αποτελεσματικότερη την υλοποίηση του δημοκρατικού συστήματο στη Γεωργία. Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Θα έχουμε τώρα μια σύντομη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαμίκινς που είναι ο εισηγητής μας για τη Γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που σας υποδεχόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Συναντηθήκαμε με την Υπουργό στην Τυφλίδα σε μια ερευνητική αποστολή στις αρχές Σεπτεμβρίου και πήγα για να διαπιστώσω η διεισόμαση τι συμβαίνει στη Γεωργία και πώς έχει κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να, να πω εισαγωγικά ότι η Γεωργία έχει μπει σε ένα μονοπάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε ακολουθήσει και η Λετωνία όταν υπέγραψε την ε, Συμφωνία Σύνδεση το 1995 και ξεκίνησε την ε, ταξιακή της πορεία. Η Γεωργία προχωρεί με ταχύς ρυθμούς και βελτιώνει και μεταρρυθμίζει το δικαστικό της σύστημα. Και παρά τις ε, διστάμενες πολιτικές απόψεις ε, που υπάρχουν στην Γεωργία, οι διεθνείς παρατηρητές έχουν αναγνωρίσει την ε, πρόοδο του δικαστικού συστήματος στη Γεωργία. Βέβαια και εγώ άκουσα αυτές τις κατηγορίες για επιλεκτική δικαιοσύνη στη Γεωργία, αλλά είναι αναφυσβήτητη και η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Γεωργία δεν είναι μια χώρα που ως διαμαγείας και χωρίς λόγο ξεκίνησε την ενταξιακή της διαδικασία. Η Γεωργία είναι μια χώρα που μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από μία εξαιτία βίωσε πόλεμο και μάλιστα η επικράτειά της είναι ακόμη διχασμένη. Εγώ, ως εισηγητής για τη Γεωργία, για τη συμφωνία αυτή και η ομάδα μου, οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες, θεωρούμε ότι η εδαφική κεραιότητα είναι μείζον ζήτημα και θα παράσχουμε την αμέριστη υποστήριξή μας προς τη Γεωργία για το θέμα αυτό. Και όταν μιλούμε για το δικαστικό σύστημα, ε, θα πρέπει και ως προς αυτό να, να, να χορηγήσουμε βοήθεια στην Γεωργία, όχι όμως μόνο στα λόγια ή να χρησιμοποιήσουμε ως πρόσχημα. Όπως είπε και η Υπουργός, ε, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στη Γεωργία. Και είναι γεγονός ότι τα δικαστήρια στη Γεωργία και οι δικαστές είναι ανεξάρτητα όσο είναι δυνατό φυσικά σε μια χώρα που εφαρμόζει, ένα, το κράτος δικαίου. Και τα κοινωνιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι παρά τις διστάμενες γνώμες που επικρατούν, που υπάρχουν μάλλον, ο γεωργιανός λαός έχει εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα της χώρας του και μάλιστα η εμπιστοσύνη αυτή αυξάνεται και ενισχύεται μήνα με το μήνα. Και η έκθεση του κυρίου Τόμας Χάμερμπερκ για την πρόοδο της Γεωργίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτή η πρόοδος να αναγνωριστεί. Σίγουρα η έκθεση βοήθησε πολύ τη Γεωργία. Και για να μην μακρηγορήσω θα ήθελα να σας ε, περιγράψω τις εμπειρίες μου. Στην Τυφλίδα είχα συνομιλίες ε, με πολλούς πολιτικούς ε, και από το κυβερνό κόμμα και από την αντιπολίτευση με εκπροσώπους ε, του κόμματος Εθνικής Ενότητας του πρώην Πρόεδρου Σακασβίλη και τους ρώτησα γιατί θεωρείτε ότι το παρόν σύστημα είναι εσφαλμένο και έχετε αντιρρήσει ως προς αυτό. Αλλά ο Σακασβίλη δεν μπόρεσε να μου δώσει απάντηση. Δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα κακό σκήμενα στο παρόν σύστημα. Ούτε είχε στοιχεία για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του ότι το σύστημα είναι προβληματικό. Και αυτή η αδυναμία του να δώσει συγκεκριμένε απαντήσεις ε, μιλάει από μόνη της. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Υπουργέ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς κυρία Υπουργέ για την ε, παρουσίασή σας ε, για την πρόοδο της γεωργίας ε, προς το ευρωπαϊκό σύστημα και την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι η σαφής άποψη του ΕΛΚ είναι ότι είμαστε πολύ καναποιημένοι με την πρόοδο που έχει ε, σημειωθεί για την ε, σφαιρική και σε βάθος Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Γεωργία και με τη συνολική διαδικασία προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την ε, ειρηνική μετάβαση σε ό,τι αφορά την εξουσία μεταξύ 2011 και 2013. Επειδή και εσεί εργαστήκατε στο Στρασβούργο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σα για την, ε, το τελευταίο ψήφισμα της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με την λειτουργία των ε, δημοκρατικών θεσμών στη Γεωργία, όπου παρά την πρόοδο που σημειώθηκε υπήρξε μια σαφή σημείωση ότι η όλη διαδικασία υποσκιάζεται από όλα τα υπόλοιπα και από την εισαγγελία και τους αξιωματούχους της προηγούμενης κυβέρνησης, το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση ε, και θέτει μάλλον ερωτήματα για τη χρήση του δικαστικού συστήματος για πολιτικούς σκόπους. Και όπως ξέρετε υπάρχει αυτή η επιλεκτική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μόνο το παράδειγμα του πρώην Πρόεδρου Σακασβίλη, αλλά και μια σειρά άλλων πολιτικών ηγετών στην Γεωργία, είναι λοιπόν βασικό για μας να κατανοήσουμε πού βρίσκεται η διαδικασία μεταρρύθμισης, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι οι μεταρρυθμίσεις που βρισκεται η διαδικασια μεταρρυθμισης προκειμενου να ειμαστε βεβαιοι οτι οι μεταρρυθμισεις που κανετε και εδώ πέρα σημειώνω την έκθεση του κυρίου Χάμερμπεργκ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτική κατάσταση όμως είναι πολύ μεταβλητή. Η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να είναι η αυριανή αντιπολίτευση. Και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε μεταβατική φάση, σε οποιαδήποτε χώρα. Το ξέρω από τη δική μου χώρα. Αυτό προαπαιτεί μια μεγάλη προσπάθεια. Σας παρακαλώ λοιπόν για σχολιάστε μου αυτό το θέμα σε σχέση με την δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μάρεκ Γιούρεκ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη αναγνώριση της ιστορίας, της 25 ης ιστορίας Γεωργίας που με πολλά προβλήματα και με ένοπλες σειράξεις ε, χτίζει έθνος. Και μετά τον ψυχρό πόλεμο ανέκτησε την ανεξαρτησία του και επειδή και εγώ κατάγομαι από μια χώρα που αντιμετώπισε παρόμοιες ε, ε, διαδικασίες γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι αυτή η δημιουργία θεσμών. Είναι δύσκολο να χτίσετε εκ του μηδενός το κράτος μετά την απελευθέρωσή σας και την ανάκτηση ανεξαρτησίας. Και φυσικά χρειάζεται ε, για κάτι τέτοιο ελάχιστη κοινωνική συνένεση. Ε, και από αυτή την άποψη μας προβληματίζουν και να ανησυχούν τα μάλα οι ειδήσει για διώξεις πρώην ε, μελών της κυβέρνησης ε, και υψηλών αξιωματούχων, όπως ε, είπε και ο προλαλής σας. Γνωρίζουμε ότι στη μετασοβιετική εποχή δύσκολο είναι να διαχωριστούν οι δημοκρατικές από τις μη δημοκρατικές δυνάμεις και η καταστολή, καταπίεσης καταπίεση βάρος ε, του πρώην Προέδρου, κατασχέσεις που γίνονται, δημεύσεις των περιουσιακών στο στοιχείο, δεν ε, δίνουν καλές εντυπώσεις για τη λειτουργία της ε, δικαιοσύνης, αλλά απλώς εκλαμβάνονται ως ανταποδοτική δικαιοσύνη ή ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών και προσωπική, και δίνει την εντύπωση προσωπικής δίωξης. Σίγουρα θέλουμε να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της Γεωργίας, αλλά από αυτή την άποψη θα πρέπει η ίδια η γεωργία να στηριχθεί σε μεγάλη κοινωνική και πολιτική συνένεση. Γιατί τέτοιες διώξεις και δράσεις θα ενοχλήσουν και θα προβληματίσουν ε, κυρίως εκείνους που ταυτίζονται περισσότερα με την προσπάθεια της γεωργίας να, να χαράξει τους θεσμούς της μετά την απόκτηση ανεξαρτησίας. Ο κύριος Αουστρεβίτσιος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Και χαιρόμαστε που ήρθατε στην Επιτροπή μας για να παρουσιάσετε την πρόοδο της Γεωργίας σε ό,τι αφορά τις δικαστικές και περαιτέρω μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Είναι σημαντικό λοιπόν να βλέπουμε ότι οι θύνοντες έχουν δυνατότητα ελεύθερη ανταλλαγής απόψεων. Ρωτώ λοιπόν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες είστε υπεύθυνοι. Διαβάζοντας τις αξιολογήσεις ε, για την ανεξαρτησία των δικαστών και του δικαστικού συστήματος και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις, αναρωτιέμαι τι γίνεται με τη νέα γενιά δικηγόρων και δικαστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο στοιχείο αυτής της νέας ε, ατμόσφαιρας αλλαγής της Γεωργίας. Σε τι βαθμό λοιπόν το δικαστικό σύστημα καλύπτεται και από νέες αρμοδιότητες, από δικαστές που έχουν φοιτήσει σε δυτικά πανεπιστήμια και επιστρέφουν στη Γεωργία για να υπηρετήσουν τη χώρα τους. Τέλος. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και η εφαρμογή έχει να κάνει με τον προπολογισμό. τι θα σχολιάζατε σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές γραμμές σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, δεδομένου δε ότι ένα τμήμα των, ε, δημοσιονομικών αυτών γραμμών προέρχεται από ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτή η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκής πλευράς πληρεί τις ανάγκες της γεωργίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκριγκούλα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μεγάλη μου τιμή που σας καλωσορίζω εδώ σήμερα. Και κυρία Πρέσβη, σας καλωσορίζω επίσης. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε εδώ σήμερα και μας εξηγείτε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα σας. Η Λετωνία πλέον, ξέρετε, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γεωργία στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, θα πρέπει να παράσχει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη με διαβουλεύσεις, με πόρους όπου αυτό χρειάζεται. Και εκ παραλλήλου θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ζώντας στην Σοβιετική Ένωση όλες οι δομές μας απήχαν παρασάγκας από τις δημοκρατικές δομές. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζητούμε από τη χώρα σας να είναι στο ίδιο επίπεδο ήδη με το επίπεδο των παλαιών δημοκρατιών. Αυτό δεν συμβαίνει σε μία νύχτα. Είναι μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Η Λετωνία λοιπόν ε, παρακολούθησε πολύ στενά τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές στη Γεωργία πριν από κάποια χρόνια και ανησυχήσαμε ιδιαίτερως με τα αποτελέσματα. Είδαμε όμως στη συνέχεια ότι υπήρξαν δημοκρατικές εκλογές πολύ καλά οργανωμένες. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι θα καταφέρετε την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είστε προς την σωστή κατεύθυνση άλλωστε. Ευθύνη δε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να παράσχει αρρωγή. Όπου αυτό χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε εκ νέου που βρίσκεστε εδώ μαζί μας, που μας μιλάτε έξω ονόματός μας. Να ξέρετε ότι είμαστε φίλοι σας και υποστηρικτές σας. Καλή σας τύχη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό. Εκτιμούμε και εμείς εδώ την παρουσία σας και τις τακτικές επαφές που έχετε με την Επιτροπή μας. Ασφαλώς, όπως επισήμεναν πολλοί συνάδελφοι και εγώ προέρχομαι από μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, είμαι από την Ουγγαρία και κατανοούμε τα προβλήματα που α, σημαίνει η οικονομική, η κοινωνική, η δικαστική μεταρρύθμιση και οι παράλληλες αυτές μεταρρυθμίσεις μεταβάσεις είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο περίπλοκο, ιδιαίτερα στη δική σας περιοχή και καλωσορίζουμε την ε, δέσμευση, τη διαρκή δέσμευση της γεωργίας στις ευρωπαϊκές αξίες και προσπαθούμε άλλωστε και εμείς τις ίδιες αξίες να προαγάγουμε στη χώρα μας και εμείς ήδη αντιμετωπίζουμε προβλήματα ενίοτε. Το μοναδικό θέμα για το οποίο θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση, παρόλο που συγχαίρω και εσάς και την κυβέρνησή σας για την εφαρμογή ενός πολύ περίπλοκου συστήματος πολιτικής μεταρρύθμισης, αν προηγουμένου σχεδόν στην περιοχή, κοινοβουλευτικές εκλογές προεδρικές, ε, προεδρική αλλαγή. Όλα αυτά εκ παραλλήλου είναι πάρα πολύ περίπλοκα σε οποιαδήποτε χώρα, πόσο μάλλον σε μια χώρα που περνάει ένα γενικό, μια γενική περίοδο μετάβασης. Σας συγχαίρω. Τονίζω όμως μία πτυχή, το οποίο, μια, η οποία βασανίζει και πλήττει όλες τις άλλες χώρες σε διαφάση μετάβασης. Κατανοούμε τον αγώνα σας κατά της διαφθοράς, και της αδιαφάνειας. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα παντού στην Ανατολική Ευρώπη, η διαφθορά. Ερωτούμε όμως, έχετε οποιαδήποτε σχέδια για να εφαρμοστεί ένα πιο στεναρό πρόγραμμα κατά της υψηλόβαθμης ε, διαφθοράς, γιατί η κοινωνία μας θεωρεί ότι αυτή η υψηλόβαθμη διαφθορά διαβρώνει την υποστήριξη στον κοινοβουλευτισμό. Έχετε λοιπόν κάποιο συνεκτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση αυτής της ε, υψηλού επίπεδου διαφθορά στη χώρα σας. Ευχαριστώ. Έχω κι εγώ μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, να τονίσω ότι για μας η Γεωργία είναι μια πολύ σημαντική χώρα και ευρύτερη ζώνη και πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το, την προμήθεια ενέργειας. Είναι κοντά στη Ρωσία και στην Τουρκία και φυσικά σημαντική δίωδος μεταφοράς ενέργειας εξαιτία και της διόδου στην Κασπία θάλασσα. Ε, είναι έκριθμη κατάσταση στην περιοχή αυτή εξαιτία και της κρίσης στην Ουκρανία. Βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη και κρίσιμη κατάσταση. Τι γίνεται με την μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας και τι κάνει η Γεωργία για να διασφαλίσει την απαραίτητη ισορροπία σε αυτή την κρίσιμη εποχή η τελευταία μιλήτρια, η κυρία Πύρη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Υπουργέ, που ήρθατε στην Επιτροπή μας και να τονίσω κάτι που και εσείς οι ίδια είπατε. Η Γεωργία έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό βήμα και στη συγκριτική αξιολόγηση με την διεξαγωγή, την ελεύθερη διεξαγωγή των εκλογών με τρόπο ανεξάρτητο. Αυτό είναι μοναδικό επιτεύγμα για όλη την γεωγραφική περιοχή και είναι κάτι που δεν ε, αντιστρέφεται στην πορεία του. Θα το θυμούνται για πάντοτε οι πολίτε τη Γεωργία και δεν αλλάζει. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει και πολλέ μεταρρυθμίσει από την προηγούμενη κυβέρνηση βεβαίω, αλλά όχι ακριβώ στο τομέα για τον οποίο είσαστε εσεί υπεύθυνοι. Νομίζω ότι για τι μεταρρυθμίσει στον δικαστικό τομέα η τελευταία κυβέρνηση άφησε πολλά ερωτηματικά. Οπότε έχετε μεγάλο φορτίο στους ώμους σας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς ε, την βιώσιμη προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, όχι απλώς να υπάρχει μια υπερψήφιση των νόμων με πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αλλά να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών και να υπάρχουν θετικές ε, συνεργασίες και με την αντιπολίτευση και τις δημοκρατικές αξίες που έχει προσφέρει. Ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα σας κύριε Υπουργέ. Λυπούμαστε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν θα είχατε την καλοσύνη λοιπόν να δώσετε τι απαντήσει και να περιοριστείτε στο δεκάλεπτο, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερως. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να σας πω ότι για να γίνω καλύτερα αντιληπτή, σε μερικές περιπτώσεις που έχω δυσκολία να εκφραστώ στα αγγλικά θα μιλήσω γαλλικά, που γνωρίζω καλύτερα. Το θέμα της επιλεκτικής δικαιοσύνης είναι κάτι που το ακούμε συχνά στην Γεωργία. Ε, αλλά όχι μόνο στη Γεωργία, αλλά και στις Βρυξέλλες ε, και από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και είναι, είναι κριτικές που ακούμε από τους φίλους μας. Και αυτά τα σχόλια έχουν ιδιαίτερη σημασία για μένα. Σημαίνει ότι οι φίλοι μας μας παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς, πολύ προσεκτικά. Και έχουν και κάποιους φόβους για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση στη χώρα μου. Και μάλιστα αυτή οι φίλοι μας, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ε, είναι οι φίλοι που βοήθησαν το λαό της Γεωργίας, όχι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και φυσικά οι φίλοι μας αυτοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνησή μου και το Υπουργείο μου εφαρμόζει την τελευταία διετία. Και οι φίλοι μας κατάλαβαν ότι οποίες από τις ε, ποινικέ ε, δίκες που εκκρεμούν στα δικαστήρια κατά υψηλό βαθμό αξιωματούχων και κατά του πρώην πρόεδρου της Γεωργίας είναι γεγονός. Στην αρχή υπήρχαν αμφιβολίες, αλλά σήμερα κανένας ε, δεν αμφισβητεί ότι στις ποινικέ αυτές υποθέσεις που εκκρεμεδικούν υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν ε, τη δικογραφία και είναι πολύ ανησυχητικά. Για παράδειγμα, την περίπτωση του πρώην Προέδρου της Γεωργίας. Για να σας δώσω μία σύντομη περιγραφή των κατηγοριών. Η ποινική υπόθεση του κυρίου Σακασφίλη αφορά την, ε, το κλείσιμο μίας, ε, ενός ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθμού και επίσης της διάλυσης με βίο τρόπο μια ειρηνικής διαδήλωσης. Θα το θυμάστε. Και επίσης τον ξηρολαδαρμό ενός, βουλευτή του κυρίου Κελαρσβίλη. Αυτές είναι οι πιο βαριές κατηγορίες που βαρύνουν τον πρώην πρόεδρο της Γεωργίας. Και μάλιστα πρόσφατα, πριν από δύο μέρες, στο Facebook, που το χρησιμοποιεί πολύ συχνά, ο κ. Σακασβίλη παραδέχτηκε ότι και ο και η κυβέρνησή του δεν κατάφεραν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας της Γεωργίας. Και αυτή η δήλωση και παραδοχή με ανακούφιση ιδιαίτερος, γιατί ε, ο λαός της Γεωργίας ε, χρειάζεται και ζητά αναγνώριση και μία παραδοχή των σφαλμάτων της προηγούμενης κυβέρνησης και του Προέδρου. Και τέτοιου είδους αναγνωρίσεις, τέτοιου είδους ομολογίες και παραδοχές και μερικές φορές ε, και το να ζητά κανείς συγγνώμη από τα θύματα θα βοηθήσουν την επανασυμφιλίωση των ομάδων της κοινωνίας στη Γεωργία. Δηλαδή των θυμάτων από τη μια πλευρά που είναι γύρω στους 20.000, είναι 20.000 τα θύματα που έχουν, ε, κατηγορεί, έχουν υποβάλει κατηγορίες και καταγγελίες ε, για άδικες δίκες, ε, κακομεταχείριση στις φυλακές, βασανιστήρια, δίμευση περιουσιών. Υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και υπάρχουν και θύματα. Κάποιος ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην επαγγελματική μου και ακαδημαϊκή μου στα και πήρα Εγώ σπούδασα στην Γαλλία, εργάστηκα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωρίζω ότι η δικαιοσύνη αφορά την ισότητα και τα δικαιώματα. Είναι αναφυσβήτητο σήμερα ότι στις ποινικέ αυτές δίκες για τις οποίες γίνεται πολλή λόγος, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, υπάρχουν γεγονότα. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι και εγώ προσωπικά και το Υπουργείο μου κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μεταρρυθμίσουμε το δικαστικό σύστημα, ώστε κάθε κατηγορούμενος ε, και ο κύριος Σακασβίλη, όταν έρθει η ώρα του, θα μπορέσουν να έχουν δίκη, δίκη στο δικαστήριο. Αυτό θα πρέπει να, να πούμε στα θύματα. Δεν μπορούμε να λέμε στα θύματα ότι ξεχάστε το, δεν πρόκειται να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Εγώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο στα θύματα, γιατί τα θύματα δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια. Και οι μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους, που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, σε περιπτώσεις που έμειναν ανεξιχνίαστες, οι μητέρες αυτές ζητούν δικαιοσύνη. Και... Ε, στην περίπτωση που έγιναν δολοφονίες από το Υπουργείο Εσωτερικών υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης ε, της εγκληματικότητας. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα και υπάρχουν στοιχεία για τις ε, κατηγορίες αυτές και τις ποινικέ διώξεις. Μερικές φορές ε, κάποιες κρίσεις αφορούν το την αντίληψη και μερικές φορές είναι και καρπός προκαταλήψεων. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις προκαταλήψεις λοιπόν. Εμείς ε, δίνουμε μάχη και εργαζόμαστε άοκνα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ε, θέλουμε την ανεξαρτησία των δικαστών και σε καμία περίπτωση να μην υπάγονται σε εκτελεστική εξουσία ούτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και φυσικά η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, του δικαστικού συστήματος προϋποθέτει μια νομοθετική μεταρρύθμιση ώστε κάθε ε, κατηγορούμενος να μπορεί να τύχει δίκης δίκης και να ε, βρίσκεται στο δικαστήριο επίσης όρης ε, απέναντι στον εισαγγελέα. Όλα αυτά είναι σημαντικά και οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν στεφθεί επιτυχία γιατί σήμερα ο Γεωργιανός δικαστής μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του μία αμφιβολία, ακόμη και όταν εκδικάζει υποθέσεις ε, υψηλόβαθμων αξιωματοχών. Γιατί στο παρελθόν ε, δεν είχε ε, δικαίωμα αμφιβολία ο δικαστής όταν εκδίκαζε υποθέσει υψηλόβαθμων αξιωματοχών. Σήμερα επιτρέπεται αυτό το δικαίωμα αμφιβολία. Και μάλιστα το... η αμφιβολία αυτή είναι ουσιαστικά στα τεκμήρια αθωότητας και ωφελεί τον κατηγορούμενο και χάρη στις μεταρρυθμίσεις έχουμε εισαγάγει αυτές τις αρχές. Οπότε με βάση το νέο σύστημα ο κάθε κατηγορούμενος ε, θα έχει δίκαιη ε, δίκη συμπεριλαμβανομένου και του πρώην Προέδρου της Γεωργίας. Μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις ή τις εσφαλμένες αντιλήψεις και μόνο έτσι θα σας δείξουμε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, ότι μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη και όλοι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην ε, δικαιοσύνη της Γεωργίας και εμπιστοσύνη στον δικαστή, το Γεωργιανό. Τώρα, για το, για το ψήφισμα ε, ε εργάστηκα για 10 χρόνια στην οργάνωση αυτή και θα μπορούσα να δουλεύω μέχρι τα 65 μου, αλλά το 2010 παρετήθηκα και επέστρεψα στη Γεωργία για να δώσω τη μάχη μου κατά της προηγούμενης κυβέρνησης εξαιτία της κατάφορης παραβίασης και μασικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτή, αυτό το ψήφισμα δείχνει ότι η γεωργιανή αντιπολίτευση έκανε τα πάντα για να υποσκάψει την εμπιστοσύνη που θα είχαν τα μέλη της ΠΑΣΕ κατά του εισηγητού και τα κατάφεραν. Και αυτό δεν είναι καθόλου θετικό για την ίδια την ΠΑΣΕ. Η η αντιπολίτευση της Γεωργίας έκανε ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των μελών της ΠΑΣΕ απέναντι στον εισηγητή της ΠΑΣΕ. Και αυτό δεν είναι καθόλου θετικό γιατί ως πρώην υπάλληλος ε, της οργάνωσης αυτής της ΠΑΣΕ ε, με ενδιαφέρει το κύρος και η έγκλη που έχει αυτή η οργάνωση στη Γεωργία. Και μάλιστα παρόμοια μέθοδο είχε χρησιμοποιήσει και η σημερινή αντιπολίτευση που ήταν κυβερνών κόμμα μεταξύ 2003 και 2012 όταν ε, επικρίθηκαν από Ευρωπαίους φίλους τους ε, αποκάλεσαν Ρώσους πράκτορες. Ο κύριος Χάμπερμπερκ που επέκρινε τότε την κυβέρνηση ε, Σακασβίλη για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων το χαρακτήρισαν ε, Ρώσο πράκτορα. Οποιοςδήποτε κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση κατηγορούνταν για κατασκοπία υπέρ των Ρώσων. Οποιαδήποτε επίκριση ή κριτική ή συμβουλή για μας είναι ανεκτήμητη σήμερα και θα την ε, αναλύσουμε επισταμένως έχουμε ένα πολύ διαφορετικό στυλ διακυβέρνησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δίμευση περιουσιών, η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, κύριε μου, ότι έχετε παραπλανηθεί και οι πληροφορίες που λάβατε είναι εσφαλμένες και ανακριβείς. Δεν εφαρμόσαμε τέτοιο μέτρο κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων ή δίμευσης περιουσιακών στοιχείων. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση για κατάσχεση ή δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε όμως μία απόφαση του Αυγούστου του 2014, μία δικαστική απόφαση που δεν θα επιχειρήσω καν να την επικρίνω. Εκεί ο Γεωργιανός δικαστής αποφάσισε να παγώσει μερικά περιουσιακά στοιχεία. Και όλοι οι δικηγόροι που είναι παρόντες θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι άλλο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και άλλο κατάσχεση δίμευση. Γιατί πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σημαίνει ότι η οικογένεια του Σακασβίλη δεν δίνεται να εκποιήσει την περιουσία της. Δεν μπορεί να κάνει πωλήσει ή άλλες δικαιοπραξίες. Και μπορώ να σας δώσω και τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει. Και Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε ο Σακασφίλη από το 2009 και μετά. Γιατί, γιατί η ποινική υπόθεση που εκκρεμωδική βάρο του αφορά περιστατικά μεταξύ 2009 και 2012. Και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσε να έχει, είχε αποκτήσει πριν το 2009 δεν περιλήθηκαν σε αυτό το πάγωμα. Έμειναν τελείως ανέγκυχτα. Οπότε όταν ε, απευθύνεται ή χρησιμοποιείτε κάποια ορολογία θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί τι όρους χρησιμοποιείτε γιατί θα πρέπει να είμαστε νομικά ακριβεί. Καμία σχέση δεν έχει το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων με την κατάσχεση ή τη δίμευση. Οι πληροφορίε που λάβατε ήταν απολύτω ανακριβεί και σφαλμένε. <laughs> Η πρέσβου μου λέει ότι θα πρέπει να ολοκληρώσω και αυτό θα ολοκληρώσω στα γαλλικά. Μίλησα για τις ε, πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι ψευδείς ή να είναι λανθασμένες όταν φτάνουν στις Βρυξέλλες ε, σε ό,τι αφορά την κυβέρνησή μας. Ε, Βεβαίω πρέπει οι πληροφορίε να συλλέγονται από πολλέ διαφορετικέ πηγέ για να είναι κανεί σίγουρο ότι έχει ενημερωθεί σωστά και να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις αποφάσει εν γνώση των γεγονότων. Όμω πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον έλεγχο των πηγών. Εμεί ω κυβέρνηση τη Γεωργία κοιτάζουμε με μάτια ανησυχία. την πορεία που ακολουθούν αυτές οι πληροφορίες, ε, όπου καμιά φορά υπάρχει μια προσπάθεια χειραγώγησης. Ε, επιστρέφω από τις ΗΠΑ, Πολιτείες, όπου ξεκινήσαμε να συζητούμε πολλά κοινά προγράμματα συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της δικαιοσύνης, και είδα εκεί ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η αντιπολίτευση σήμερα, ετοιμάζονται να δημιουργήσουν παράλληλες δομές με τις, ε, του κράτους. Δηλαδή παράλληλες ε, πρεσβείες ας πούμε που θα τις ονομάσουν think tank και ε, επίσης και άλλες υπηρεσίες για να αποδείξουν ότι η Γεωργία ε, είναι στον κακό δρόμο. Η Γεωργία δεν έχει πάρει τον κακό δρόμο, το αρνούμε αυτό. Αυτό που χρειάζεται η Γεωργία είναι η διαρκή σας στήριξη, η προσοχή που θα δίνετε σε κάθε μια από τις δράσεις μας και το Συμβούλιο. Μάλλον η Συμβουλή σας. Είναι πολύτιμες οι συμβουλές σας, ε, διότι οι συμβουλές του εισηγητή, ε, του κυρίου Χάμεμπεργκ, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δικές σας, είναι πολύτιμες όλα αυτά τα χρόνια. Μας βοηθούν να ακολουθούμε το σωστό δρόμο. Και πάλι σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε και που δεχτήκατε να με ακούσετε. Βεβαίως δεν μπόρεσα να σας προσφέρω όλες τις πληροφορίες που θα ήθελα, διότι τα θέματα είναι ιδιαίτερα είναι ευρέα. και υπήρχαν πολλές ειδικέ λεπτομέρειες νομικές που θα έπρεπε να εξηγήσει κανείς, αλλά ό,τι περαιτέρω πληροφορία χρειάζεστε για τις μεταρρυθμίσεις μας και για την ανοικοδόμηση του κράτους, στην οποία συμμετέχω με τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης, ευχαρίστω να σας τις δώσω. Έχουμε έναν κοινό στόχο, έναν και μοναδικό. Δεν υπάρχουν άλλοι. Να μην παραμείνουμε πάρα πολύ καιρό στην εξουσία, προκειμένου να μην ξεχάσουμε ότι και δημοκρατία υπάρχει μόνο όταν υπάρχει αναλλαγή. Ίσως η σημερινή αντιπολίτευση να επανέλθει στην κυβέρνηση το 2016. Θέλουμε λοιπόν να οικοδομηθεί ένα κράτος που να έχει υποδομές, να έχει ε, δομές που να λειτουργούν και δεν θα θέλα ποτέ ξανά η γεωργία ως κράτος να εξαρτάται από πρόσωπα και προσωπικότητες. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Θέλουμε τη θεσμική δημοκρατία για τη γεωργία και αυτό προσωπικώς επιθυμώ και εγώ και η κυβέρνησή μου. Και ε, υπολογίζουμε στη διαρκή σας στήριξη. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ πιστεύω ακράδαντα ότι οι σχέσεις ε, με, τους, με τις γειτονικές χώρες, ε, ακόμη και με τη Ρωσία, μπορούν να είναι συμβατές ε, με τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις για να ασφαλίσετε τη σταθερότητα και την κυριαρχία της Γεωργίας σε ένα θέμα που ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας στο σπίτι σας μπορείτε να έρχεστε όποτε το επιθυμείτε. Ενός λεπτού διακοπή και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση λίγο αργότερα. Le voy a dar la palabra ahora si quiere intervenir al señor Maminkins. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαμίνκης τώρα, αν θέλει να προσθέσει κάτι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή, την προσοχή στο σχέδιο έκθεσης για την ετοιμότητα της ε, γεωργίας σε ό,τι αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας. Ε, συμμετείχα σε μια διερευνητική αποστολή στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου στην ε, Γεωργία και είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με όλους σχεδόν. Ε, με εκπροσώπου τη κυβέρνηση, τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τον υπουργό εξωτερικών, ε, δικαιοσύνη και με μη κυβερνητικέ οργανώσει με την αντιπολίτευση, εκπροσώπου σεξουαλικών ε, μειονοτήτων, εκπροσώπου οργανώσεων θρησκευτικού υπόβαθρου τη Ορθόδοξη Εκκλησία, όπω όλοι ξέρουμε, η Εκκλησία έχει σημαντικό αντίκτυπο στις διαδικασίες αυτές με 95% των Γεωργιανών να εκφράζουν εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Διαπίστωσα επίσης ε, τα παράνομα σύνορα μεταξύ στην Ενώτιο Σωτία. Ένα τμήμα των σύνορων το οποίο έχει κατασκευαστεί παράνομα. Είναι αδύνατον να το περάσει κανείς, σωματικά αδύνατον. Και αυτό προκαλεί προβλήματα, για παράδειγμα, στις συντάξεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι, κατά τη γνώμη μου, η μελλοντική απελευθέρωση από το καθεστώς θεωρήσεων στη Γεωργία θα βοηθήσει εν μέρη να επιληθεί το ζήτημα της εδάφικης ακαιρεότητας, γιατί όσοι ζουν στην Αμπχαζία στην Νότια Οσοτία σήμερα, θα είχαν με τον τρόπο αυτό την ευκαιρία να επιστρέψουν στο γεωργιανό τους διαβατήριο και να επανενταχθούν στην γεωργία. Να εκφράσω λοιπόν την ευγνωμοσύνη μου στους κοιόδης εισηγητές με τους οποίους ήδη είχα την ευκαιρία να συναντηθώ από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και με όσους θα συναντήσω τους επόμενες ημέρες και προσβλέπω και στα κριτικά σας σχόλια ασφαλώς. Ο κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Εκτιμώ ιδιαίτερος ε, που μπήκατε στον κόπο να μεταβείτε και στη Γεωργία αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και να δείτε ιδίως την κατάσταση στη Γεωργία. Φάνηκε άλλωστε και στα σχόλια που κάνατε μετά την παρέμβαση της ε, Υπουργού ε, Τσουλουκιάνη. Και στα πλαίσια τη Συμφωνία Σύνδεση, αλλά και στα πλαίσια τη Φερική ε, και σε βάθο Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, θα ήθελα να πω ότι εμεί είμαστε υπέρ ε, τη κύρωση και υπέρ τη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δύο συμφωνιών και τη Συμφωνία Σύνδεση και τη Φερική και σε βάθο Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και οι δύο συμφωνίε στην Γεωργία να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές αυτή την δύσκολη μεταβατική κατάσταση που βρίσκεται. Και σίγουρα η προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να επισκιαστεί από την κρίση στην Ουκρανία. Ε, και, και για την ε, Μολδαβία θα πρέπει να θετήσουμε την, την ίδια προοπτική, το ίδιο πρίσμα. Στην ε, χώρα μου θα υιοθετήσουμε ταυτόχρονα και τις τρεις συμφωνίες ε, και τις συμφωνίες είδης και τη σφαιρική και σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Επέμεινα μάλιστα να γίνει αυτό, αυτή η έγκριση ταυτόχρονα και όσο πιο εύρυθμα γίνεται. Και όταν εξετάζουμε την ε, συνολική αξιολόγηση, ιδιαίτερα και μετά την ενημέρωση που μας έκανε η Υπουργός Δικαιοσύνης της Γεωργίας, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς το περιεχόμενο και του δικού μας ψηφίσματος. Αναφέρθηκε το πρόσφατο ψήφισμα για την κατάσταση ε, της δικαιοσύνης και την πορεία των μεταρρυθμίσεων από την ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα πρέπει οι εξουσίες της κυβέρνησης να μην χρησιμοποιηθούν εις βάρος της αντιπολίτευσης. Γιατί κάτι τέτοιο δεν συμβάλλει στην δημοκρατική ανάπτυξη της Γεωργίας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά και κατά την υποβολή των τροπολογιών μας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθεί, θα ενισχυθεί το δικαστικό σύστημα προκειμένου να αποφευθεί η πολιτική ανταπόδοση, η εκδίκηση και να εξασφαλιστούν δίκαιες δίκες. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και αναφέρθηκαν από πολλούς ομιλητές. Θέλουμε μια θετική ευρωπαϊκή προοπτική της γεωργίας και μια στιβαρή δημοκρατία που θα λειτουργεί εύρυθμα. Αυτή είναι η στόχη νομίζω όλων μας για τη γεωργία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκριγκούλε. Um, um, Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Αφού διάβασα το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Μαμίκινς, πρέπει να πω ότι κατά την άποψή μας είναι πολύ καλό το σχέδιο, πολύ καλό το κείμενο, πολύ αντικειμενικό, αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης και είναι πολύ ευχάριστο που ο εισηγητής έχει επισκεφτεί τη χώρα, έχει συναντήσει πολιτικούς από όλο το πολιτικό φάσμα και εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ως ε, νέα ευρωβουλευτής θέλω να ευχηθώ στον κύριο Μαμίκινς να συνεχίσει τη δουλειά του στην έκθεση αυτή και να ολοκληρωθεί η έκθεση για την Γεωργία όπως πέτυχε αντιστοίχως και η επεξεργασία της συμφωνίας με τη Μολδαβία. Ο κύριος Μιζηρίξ, ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την καλή του δουλειά. Είναι πάρα πολύ συνεκτική και την ε, προετοίμασε πάρα πολύ γρήγορα. Πάντα πολύ σημαντικό αυτό στην Επιτροπή μας. Γενικά συμφωνούμε με τις περισσότερες δηλώσεις. Θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες οι οποίες το πλήστον δεν άπτονται του πυρήνα της έκθεσης. Θα ήθελα παρά, παρόλα αυτά να αναφερθώ σε δύο ζητήματα τα οποία και σκοπεύουμε να τονίσουμε με την ε, σε βάθος συμφωνία και με την συμμετοχή της Γεωργίας στον ΠΟΕ θέλουμε να διασφαλίσουμε και ως Επιτροπή ότι η Γεωργία δεν θα στρεβλώσει τις εμπορικές της σχέσεις με την υπόλοιπη περιφέρεια. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν τη Γεωργία αλλά διατηρώντας παράλληλα τις σχέσεις που έχει στην περιοχή. Αυτό και οικονομικός αλλά και πολιτικός. Πώς είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που κάπως θεωρούμε ότι λείπει από την έκθεση είναι η αντίποτε αναφορά στις ε, συζητήσεις στη Γενέβη. Σίγουρα το θέμα της γεωργίας θα πρέπει να αναφέρεται και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, όχι μόνο σε επίπεδο διπλωματίας. Και Επίσης υπάρχουν και κάποιες επενδύσεις ενεργειακής πολιτικής στο νότο της Γεωργίας, κυρίως υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που εξ γνωρίζουμε δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστήμω λοιπόν την προσοχή της ε, Επιτροπής ότι ενδεχομένως εδώ να χρειάζεται πλήρη συμμόρφωση με τα επίπεδα που προβλέπει η νομοθεσία πρωτού τεθούν σε εφαρμογή και σε λειτουργία. Κατά τα άλλα όμως είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την έκθεση. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο για ένα-δύο μιλητέ. πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή μας για να ολοκληρώσει. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, πολύ ευχαρίστω. Αλλιώς θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Μαμίκιν, στον εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ και πάλι, συνάδελφοι για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας θα τα λάβω υπόψη. Η προθεσμία και κατάθεση τροπολογιών, όπως βλέπετε στην ατζέντα, είναι 22 Σεπτεμβρίου. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους όσοι ενδιαφερθήκατε και διαβάσατε την έκθεση και ανταλλάξατε τις απόψεις σας μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για να αλλάξει ο πρόεδρος και να έρθει και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, αναλαμβάνω εγώ τώρα την Προεδρία της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή γι' αυτό και καλωσορίζω εγκάρδια τον ε, Υπουργό Βόλκαν Μποσκύρ, που είναι Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και επικεφαλής διαπραγμάτευσης ε, της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι γνωστός εκεί ο πρόσωπο, είτε από την προηγούμενη διπλωματική του σταδιοδρομία, είτε από την ιδιότητά τους βουλευτή της ε, Τουρκικής ε, Εθνοσυνέλευσης και ήταν και πρόεδρος άλλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ήταν και μόνιμος αντιπρόσωπος ε, της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικός γραμματέας ή υφυπουργός της Τουρκίας πριν να λάβει το Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας. Έρχεται για συζήτηση μετά την τελευταία συζήτηση με τον Στέφαν Φίλε, τον αρμόδιο για τη διεύρυνση επίτροπο, μετά την πρόσφατη έκθεση πρώτα της 8ης Οκτωβρίου για την Τουρκία και θα συζητήσουμε την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με, της Τουρκίας καθώς και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας θα προχωρήσει μόνο με βάση την υλοποίηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων και προς το αμοιβαίο όφελος. Γνωρίζετε ότι όπως και η Τουρκία, η πατρίδα μου ξεκίνησε την διαδικασία αυτή στις 3 Οκτωβρίου του 2005 στο Λουξεμβούργο και είδαμε ότι η δυναμική και εξέλιξη αυτής της ενταξιακής διαδικασίας είναι πολύ πιο περίπλοκη και πολύ πιο απαιτητική στη δική σας περίπτωση από ό,τι ήταν στην περίπτωση της Κροατίας. Είναι, κάθε ενταξιακή διαδικασία είναι μοναδική και ε, έχουμε πολλά χρόνια που έχουν περάσει από την ε, σύναψη της Συμφωνίας Είδησης ε, με την Άγκυρα. Θα μας ενημερώσετε λοιπόν για την πορεία των μεταρρυθμίσεων σε θέματα δικαστικά και θεμελιωδών ελευθεριών και επίσης θα μας εξηγήσετε την ευθυγράμμιση της εξωτερικής τουρκικής πολιτικής με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό θέμα γιατί βρίσκεται, βρίσκεται σε μια πολύ απαιτητική περιοχή με τεράστιες προκλήσεις. Βέβαια κάθε χώρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά ειδικά λόγω της κρίσης ε, στο Ιράκ στη Συρία η χώρα σας βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη ζώνη. Έχουμε επίσης το θέμα της ε, καταπολέμησης του ISIS και το κουρδικό σύστημα, αλλά και το κουρδικό πρόβλημα στα σύνορα της Τουρκίας, ιδιαίτερα στην πόλη Κομπάνη. Θα σας δώσω το λόγο κύριε Υπουργέ για 10 με 15 λεπτά και παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη συζήτηση να το δηλώσουν. Ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Βλέπω πολλά πρόσωπα υπό την προηγούμενη ιδιότητά μου και επίσης πολλά, που τα θυμάμαι την προηγούμενη μου ιδιότητα και πολλά νέα μέλη σε αυτή την Επιτροπή. Είναι χαρά να βρίσκεται εδώ οποιοδήποτε χρειάζεται να εκφωνήσει μια ομιλία εδώ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θα μιλήσω για τις σκέψεις της Τουρκίας ή τέλος πάντων την νέα στρατηγική της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι σκοπεύουμε να κάνουμε για να μην υπάρχει ένας μονόλογος αλλά ένας νέος διάλογος μεταξύ μας. Με τα χαρά θα ακούσω λοιπόν τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρώτα απ' όλα στην Τουρκία ξεκινά μια νέα εποχή ο Τούρκος πρόεδρος για πρώτη φορά εξελέγει απευθείας άμεσα. Έχουμε ένα νέο πρόεδρο, ένα νέο πρωθυπουργό και νέα κυβέρνηση. Όταν το συζητούμε μεταξύ μας μιλάμε για μια νέα Τουρκία. Βλέπετε να εφαρμόζονται νέες προσεγγίσεις ή να επανεπιβεβαιώνονται κάποιες από τις προηγούμενες νέες αποφάσεις με έντονο τρόπο κιόλα και με αποφασιστικότητα ιδίως ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα μέτρα αυτά αφορούσε τις διπλωματικέ υπηρεσίες. Και νομίζω ότι έχει νόημα το τι μεγάλη επένδυση έχει γίνει από την πλευρά των διπλωματικών μας υπηρεσιών για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε εκλογές λοιπόν, ε, νέα βουλή, κάποια πρόσωπα απεχώρησαν, αλλά πολλοί από τους εναπομείναντες είναι και πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι να ε, συμμετάσχουν στην διαδικασία έλεξη αποφάσεων ε, το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια νέα επιτροπή, νέο πρόεδρο του Συμβουλίου, νέο κοινοβούλιο, νέα Ευρώπη λοιπόν, αλλά και νέα Τουρκία. Μεγάλη σύμπτωση την ίδια χρονική στιγμή. Νομίζω θα πρέπει αυτήν την ε, συγκυρία να την εκμεταλλευτούμε ε, για να εξυπηρετήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Να εξηγήσω ότι έχουμε κάνει πρόσφατα λοιπόν Πρώτα απ' όλα έχουμε χαράξει και έχουμε εκπονήσει μια νέα στατηγική για τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω διανύμει το σχετικό έγγραφο, ελπίζω ότι το έχετε διαβάσει. Αλλά θα είναι τρόπον τεινά το σύνταγμα που θα καθορίσει την ε, πρόοδο των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εφ' εξής. Αυτή θα είναι η βασική πλατφόρμα το εφαλτήριο από το οποίο θα λειτουργήσει η διαμόρφωση των, σχέσεων, των μας. Έπειτα υπάρχουν τρεις πυλώνες. Πρώτα απ' όλα οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Η Τουρκία μεγάλη έμφαση δίνει κυρίως στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και Αυτό ίσχυε και όταν ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλεγε ότι η Τουρκία εκπλήρωνε επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια. Βέβαια, η απόσταση μεταξύ του ε, πληρεί επαρκώς ή πλήρως, καλύπτει πλήρως, είναι ακόμα μια απόσταση που πρέπει να διανύσουμε. Θα πρέπει λοιπόν οι υπουργοί μα ε, δικαιοσύνη εξωτερικών υποθέσεων και για, την Ευρωπαϊκή, για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώ να συναντηθούν, αλλά να ετοιμάσουν και σχετικές δηλώσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις να εκπονηθούν, να προγραμματιστούν, να υλοποιηθούν. Α, τη Δευτέρα α, ζήτησα από το Υπουργικό Συμβούλιο να αλλάξει τον τίτλο της ομάδας εργασίας που υπάρχει από το 2004, μάλλον τρία ε, για τις μεταρρυθμίσεις, ε, σε ομάδα δράσης για τις μεταρρυθμίσεις και όχι ομάδα ε, μελέτης για τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, κάτι άλλο που είναι καθοριστική σημασία για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρόγραμμα για την ε, πρόοδο των σχέσεών μας. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα δράσης υπόψη σε δύο φάσεις. Το πρώτο προβλέπει ε, πρωτογενή νομοθεσία και ένα χρονοδιάγραμμα ε, για το διάστημα ως το 2015 και μετά για το διάστημα 2015-2019. Το πρώτο τμήμα είναι ήδη έτοιμο, το ενέκρινε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σήμερα το παρουσίασα στην ε, Υπηρεσία Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιμένω και τη δική τους αποτίμηση και τις δικές τους συνεισφορές ε, εντός του μήνα ε, Οκτωβρίου. Το επόμενο τμήμα θα ακολουθήσει στα μέσα Νοεμβρίου και επίσης θα το κοινοποιήσουμε αμέσως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Νοέμβρη. Για αυτά τα πολύ σημαντικά βήματα, τα δύο αυτά σημαντικά βήματα πρόοδου, έχουμε και μια ε, εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, ο οποίος προβλέπει θεσμικά σε επίπεδο Υπουργείων της Τουρκίας ώστε να συνεργάζονται με τους ομολόγους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποτε υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση νομοσχεδίου, οποιοδήποτε νομοθετική κίνηση θα υπάρχει έλεγχος για να δούμε κατά πόσον αυτά συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο αλλά και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το τρίτο σημείο. Ο τρίτος πυλώνας είναι η επικοινωνιακή μας στρατηγική. Έχει ήδη ετοιμαστεί και έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση και σήμερα σε συνέντευξη τύπου στις 4 ε, θα την παρουσιάσω και επισήμως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η τουρκική επικοινωνιακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες φορές η εικόνα που έχουμε είναι ε, σφαλμένη διότι ε, στις συζητήσει μας πολλές φορές επειδή δεν έχουμε εξηγήσει αρκετά τις έννοιες όπως τις καταλαβαίνουμε η μεν και οι δε έχουν προκύψει κάποιες παρανοήσεις θέλουμε λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος που ε, αντιμετωπίζουν την Τουρκία τα ευρωπαϊκά κράτη Θέλουμε να αλλάξει αυτή η εικόνα ε, για να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει ε, χάσει ένα μέρος από το κύριο της στην Τουρκία. Έχει αλλάξει η εικόνα της. Σκέφτονται ας πούμε στην Τουρκία οι άνθρωποι γιατί τη θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μας χρειάζεται. Έχει αρκετό πλούτο. Μπορεί να βοηθήσει... Εδώ δεν μπορεί να βοηθήσει χώρες που έχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί στραβές ε, αντιλήψεις που έχουν ριζώσει η στατηγική μας σκοπό έχει να αποκαταστήσουμε την εικόνα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστρόφως. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών, διότι στην αρχή της δεκαετίας του 80 είχαμε λιγότερες από 20 ενώσεις των πολιτών, είναι κυβερνητικές οργανώσεις, τώρα έχουμε περισσότερες από 1900. 19.000 μάλλον και ίσως και πάνω από 20.000 συλλόγους, ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Είναι τεράστιο αυτό για μια δημοκρατική χώρα ως αριθμός ε, και δεν μπορώ να φανταστώ και άλλο τρόπο για να λειτουργεί από δημοκρατική σκοπιά εύρυθμα μια οποιαδήποτε χώρα. Είναι σημαντική παρουσία των οργανώσεων αυτών λοιπόν και θα είναι μέρος της επικοινωνικής μας πολιτικής για να εξηγήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία το τι ε, σκέφτονται οι ΜΕΝ και οι ΔΕ, αλλά και να βοηθήσουν στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που σας ανέφερα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας βεβαίως είναι εξίσου σημαντικός, τα προγράμματα αυτά που ανέφερα. Ωστόσο ε, να μην υπάρχουν ε, αντιφάσεις προς τους νόμους, τα νομοσχέδια που ετοιμάζονται. Έτσι, οι άπαντες θα μπορούν να δουν τι ε, προγραμματίζει η Τουρκία ως το 2015 και μετά και ως το 2019. Αυτό είναι σημαντικό και για τη δική μας την νομοθετική πειθαρχία και για να ασκήσουμε και πίεση, εφόσον όλα αυτά θα βρίσκονται επί χάρτου, να ασκήσουμε πίεση αλλά και να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ε, για το ποια μέτρα είναι προτεραιότητας και αναγκαία και ποια δεν έχουν περιληφθεί ενδεχομένως στο πρόγραμμα και για ποιο λόγο. Θα πρέπει επίσης να επικρατήσει ένα νέο ύφο. συμμετείχα σε συνεδριάσεις αυτής της σημαντικότατης επιτροπής ή της κοινής της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πια ένα νέο ύφος, ε, ένα νέο κλίμα στις σχέσεις μας. Να ακούμε μεν τους δε, να επικρίνουμε μεν τους δε, να σεβόμαστε τις επικρίσεις που μπορεί να εκφράζονται αμοιβαίως και να δημιουργηθεί μια νέα ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης. Ίσως κάποιες προηγούμενες συνεδριάσεις να κατέληγαν όχι απλώς σε μη θετικά αποτέλεσμα, αλλά σε κάποιες ζημινιές. Αυτό θα θέλαμε να αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν να επικρατήσει ένα νέο υφός και θα κάνω ό,τι μπορώ για να το επιβάλλω, ώστε να είναι ωφέλιμες οι συνεδριάσεις επικοδομητικέ και να μην έχουν αντίστροφα από επιθυμητά αποτελέσματα. Με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω, να σας δώσω το χρόνο για ερωτήσεις, ώστε να ξεκινήσει όντως να πάρει σάρκα και ε, ο διάλογος. Επίσης βλέπω εδώ τη νέα σας εισηγήτρια, της εύχομαι καλή τύχη. Θα μιλήσουμε σύντομα για κατηδίαν και εύχομαι να έχουμε μια άριστη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε Υπουργέ τηρήσατε και τα χρονικά όρια. Προκειμένου λοιπόν να διοργανώσουμε κάπως τη συζήτησή μας, να την οργανώσουμε και τις παρεμβάσεις σας, θα δώσω πρώτο το λόγο στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ε, ε Αντιπροσωπείας στην Τουρκία και μετά στην εισηγήτρια και στον κύριο ε, Σκιώδη εισηγητή, τον κύριο Φανόρτεν, ο οποίος όμως είχε, έφυγε ζητά συγγνώμη για την ε, απουσία του και κύριε Κεφαλογιάννη λοιπόν έχετε το λόγο. Sorry. Sorry. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας. Ε, προσβλέπουμε σε μια ως Επιτροπή, Κοινή, Ευρωπαϊκή, Κοινή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας προσβλέπουμε σε μια άριστη συνεργασία μαζί του η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εταίρος της Τουρκίας. Ε, οι διαδικασίες ε, ε, για την Τουρκία δεν έχουν προχωρήσει όπως πρέπει. Εμείς έχουμε την διάθεση το επόμενο διάστημα που θα ακολουθήσει σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας από το Κοινοβούλιο στην Τουρκία να κάνουμε βήματα θετικά. Βεβαίως πάντα κάτω από το πρίσμα των αρχών και των κεκτημένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να διευθετήσουμε με την Τουρκία. Πιστεύουμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία εγγυάται τη σταθερότητα στην περιοχή αλλά χρειάζεται να υπάρχουν κανόνες ε, καλής γειτονίας με όλες τις χώρες της περιοχής και θα ήθελα να ε, κάνω και μία ερώτηση στον κύριο Υπουργό κατά πόσον και με αφορμή τα τελευταία θέματα που έχουν προκύψει στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κατά πόσον η Τουρκία είναι έτοιμη να ε, υιοθετήσει τις συμφωνίες ε, των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης και ποια είναι η θέση της Τουρκίας για την αποκλειστική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κύπρου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ κύριε Κεφαλαγιάννη, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάκη Χατζηγεργίου. Κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Είμαι ο Τάκης Χατζηγεωργίου, είμαι ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ από την Κύπρο. Θέλω καταρχήν να σας πω ότι ε, παρακολουθώ μια μετριοπαθή στάση, ιδιαίτερα εκ μέρους ημών, ε, όσον αφορά θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι που πρέπει να, να το υπογραμμίσω. Ε, θέλω όμως να συμφωνήσω επίσης μαζί σας σε κάποιες δηλώσεις που έχετε κάνει παλαιότερα και έρχομαι σιγά σιγά στο Κυπριακό ότι υπάρχουν χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες ουσιαστικά κρύβονται πίσω από το Κυπριακό για να εμποδίσουν την ένταξη της Τουρκίας. Υπάρχουν μάλιστα δηλώσεις του τύπου δεν εντάσσεται η Τουρκία αν δεν λυθεί το Κυπριακό που ενώ ακούγεται πάρα πολύ ωραία δήλωση στην πραγματικότητα μπορεί να σημαίνει ας μην ενταχθεί ποτέ η Τουρκία και ας μην λυθεί ποτέ το Κυπριακό. Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι για να ξεμπροστιαστούν οι χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν ε, αυτό το πρόβλημα. Όμως νομίζω ότι στην προσπάθειά σας να ενταχθείτε πρέπει να αναζητήσετε πραγματικούς συμμάχους και τους πραγματικούς συμμάχους θα τους βρείτε μόνο στους εκπροσώπους της Κύπρου και της Ελλάδας και κάποιων άλλων χωρών. Άρα πρέπει να στραφείτε στη συνεργασία, στη συνέργεια κοινών συμφερόντων προς την ίδια κατεύθυνση. Και ενώ επιθυμείτε εσείς και ασφαλώς εργάζονται και πάρα πολλοί άλλοι μέσα στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή για να ανοίξουν κεφάλαια. Δυστυχώς όσο και αν ενοχλεί το να αγνοεί κάποιος ότι η κύρια αιτία του μη ανοίγματος των κεφαλαίων είναι το το κυπριακό, είναι σαν να αποφεύγει κανείς να δει τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο. Πρέπει να στραφείτε ξανά προς την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Και νομίζω ότι οι ενέργειες οι τελευταίες της χώρας σας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου είναι επιζήμιες, παραβλάπτουν πάρα πολύ τη διαδικασία της επίλυσης. Ήδη υπάρχει αναστολή συμμετοχής στις ε, συνομιλίες από τον πρόεδρο της Κύπρου και κλείνω με μια ερώτηση που αφορά ευρύτερα ζητήματα και αφορά το Ισλαμικό κράτος και την επίθεσή του ενάντια στους Κούρδους της περιοχής. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα συνεχίσετε να έχετε την ίδια στάση μη ουσιαστική συμμετοχή ε, ενάντια στην, ε, στο Ισλαμικό κράτος διότι επιθυμείτε την ταυτόχρονη πτώση ε, του καθεστώτος του Άσαντ ή θα επιχειρήσετε κάποια στιγμή μια μεταστροφή πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χατζηγεωργίου και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον, στην εισηγητρία μας, την κυρία Πύρη και μετά στον Σκιώδη, την κύριε Σε Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημερωτική παρουσίασή σας αυτή. Είναι σαφές ότι και εσείς και η ομάδα σας είστε δεσμευμένοι σε ό,τι αφορά την διαδικασία προσχώρησης και στη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προετοιμάσατε τονίζετε ότι θα συνεχίσετε την αρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το καλωσορίζουμε αυτό και θεωρούμε ότι αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα. Ότι η Τουρκία δεσμεύεται να συνεχίσει τη δουλειά στον τομέα του κράτους δικαίου και δημοκρατισμού και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ελήψη επίσημων διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια 23 και 24 αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ιδανική η κατάσταση. Και εδώ πέρα στην έκθεση Women Rights που εγκρίθηκε πέρσι ε, ζητήσαμε να, να γίνει τη διαδικασία ελέγχου των κεφαλαίων αυτών. Καλωσορίζουμε λοιπόν τις συζητήσεις παρά το μπλοκ που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Θέλουμε όμως να υπάρχει και εναρμόνιση με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουν τονιστεί κάποιες θετικέ εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ζητήματα που έχουν επισημαθεί όμως και ζητήματα τα οποία είναι ενσυχητικά σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Δύο θέματα θα ήθελα να θέσω. Το παλιό γνωστό θέμα, η ανεξαρτησία του δικαστικού, η, ο διαχωρισμός των ε, εκτελεστικών εξουσιών και του ε, νομοθετικού σκέλους. Και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σα σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να σας έχω την ευκαιρία να σας καλωσορίζω και στο μέλλον και προσβλέπουμε σε μια καρποφόρα συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Μαξιγκαλός. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Αν θα θέλετε λοιπόν να βάλετε τα ακουστικά σας. Εγώ λοιπόν είμαι από την Σουηδία και ήμουνα επί 8 χρόνια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της, του Συνδικού Κοινοβουλίου και η Σουηδία είναι ίσως ένας από τους μεγαλύτερους υπέρμαχους της προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο το πολιτικό φάσμα από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά του πολιτικού φάσματος υπάρχει ευρεία υποστήριξη υπέρ της προσχώρησης της Τουρκίας και συχνά αναφέρουμε αυτό που ανέφερε και ο Υπουργό ότι πρέπει να ακούμε και να μπορούμε να ασκούμε κριτική γιατί οι καλοί φίλοι σχολιάζουν και τα καλώς και τα κακώς κείμενα. Εδώ εκπροσωπώ την ομάδα των Πρασίνων και βλέπουμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό θέμα το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερο σήμερα είναι η κατάσταση στο κομπάνι. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε πιο πολλά για το πώς ε, θεωρεί η Τουρκία ότι διαμορφώνεται ο ρόλος που πρέπει να διδραματίσει εκεί. Και βλέπουμε διαρκώς ότι υπάρχουν ε, ενδείξεις όχι μόνο από Κούρδους αλλά και από άλλες πλευρές ότι η Τουρκία ουσιαστικά αποτρέπει την άμυνα των ε, Κούρδων αντί να τη διευκολύνει. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούμε με τους Τουρκούς στο θέμα αυτό προκειμένου να υποχωρήσει η οργάνωση ίσης. Δεν είναι μόνο ο Ασάντ εχθρός ε, της Συρίας, είναι και το ίσης. Και ίσως λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Κάτι τώρα που μας ανησυχεί περαιτέρω η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της Τουρκίας και των ανταρτών του ΠΚΚ. Ξέρουμε ότι συνεχίζονται συζητήσεις εδώ και κάποιο καιρό και θέλουμε να μας διαβεβαιώσετε ότι οι συζητήσεις αυτές δεν είναι απλά μόστρα. Ότι πραγματικά διεξαγάγονται και όχι μόνο για να δείξουν ε, σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι α, γίνονται διαπραγματεύσει και γίνονται συζητήσεις. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει ένα περιεχόμενο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα για τι επιθέσει αυτέ κατά των Κουρδών. Ένα περαιτέρω θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και το οποίο έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια είναι το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας έκφρασης. Ζητήματα που μας ανησυχούν και θα θέλαμε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σεβάιος. Θα πρότεινα να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων και κατόπιν θα ακούσουμε τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Πρώτα την κυρία Λίο Μαρή, μετά τον κύριο Παντζέρη, τον κύριο Τάνοκ, τον Σάκε, Βερζιά, τον κύριο Πιτίδιο, τον κύριο Μαυρίδη και άλλοι. Παρακαλώ θέλει κανείς άλλο το λόγο να το δηλώσει και να μην ξεπεράσουν οι ομιλητές το ένα με 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους που μιλήσαν, τους εκπροσώπους των επιτροπών, τον, την εισηγήτρια, τους εκπροσώπους κάποιων ομάδων, το σκιώδη εισηγητή. Ξέχασα να συγχαρώ τον κύριο Κεφαλογιάννη που είναι πλέον συμπρόεδρος της JPC. Θα συναντηθούμε και προσωπικά αργότερα και αδειμονώ για την ιδιωτική συνομιλία που θα έχουμε και φυσικά θα συζητήσουμε μαζί κύριε Κεφαλογιάννη για να δούμε πώς θα κάνουμε αυτή την JPC που υπάρχει από το 1966 και συστήθηκε ως πλατφόρμα για να διευκολύνει τις σχέσεις, όχι να τις παρεμποδίσει ή να τις παραβλάψει. Οπότε θα έχω συζήτηση με τον αγαπητό, το φίλο, το συνάδελφο, να δούμε νέες μεθοδολογίες για να πραγματώσουμε αυτή τη φιλοδοξία. Και φυσικά θα ήθελα να, είστε ως, να δράσετε ως διαιτητής. Και εγώ ήμουν, το πάλι ποτέ πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα να είστε δίκαιος απέναντι σε όλες τις απόψεις που θα ακουστούν στην Επιτροπή. Και είμαι βέβαιος ότι με τις ικανότητες που έχετε θα καταφέρετε να διαδραματίσετε αυτό το ρόλο. Θα ήθελα τώρα κάπως να ομαδοποιήσω τα ερωτήματα και να σας εξηγήσω τη θέση μου για τα επιμέρους ζητήματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με, τις, καταστάσεις, με την κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ, στα νότια μας σύνορα. Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα και την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο και φυσικά και την Τουρκία. Και φυσικά είναι και προτεραιότητα της Επιτροπής Εξωτερικών. Στη Γερμανία έλαβα μέρος στην ευρίαση της αντίστοιχη επιτροπής και φυσικά ανέκυψαν τα ίδια ερωτήματα. οι τελευταίες εξελίξεις ε, στη Συρία και το Ιράκ έχουν σχέση με την δημιουργία αυτής της περίεργης οντότητας, αυτής της τρομοκρατικής ε, οργάνωσης που κατά κάποιο τρόπο μας ευνηδίασε όλους, γιατί έχει μια νέα νοοτροπία, έχει ένα νέο στυλ, ένα νέο τρόπο να σκοτώνει ανθρώπους και η οργάνωση αυτή μπήκε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας ε, με μια νέα μορφή τρομοκρατίας. Πρόκειται για μια νέα τρομοκρατική οργάνωση και δεν καταφέραμε να δώσουμε μια στιβαρή απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Αυτό αποκαλείται η οργάνωση αυτή Ισλαμικό κράτος. Μερικοί του ε, ε, ονομάζουν Ισίλ, το Έλληνε Λεβάντε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνος χαρακτηρισμός, γιατί το Λεβάντε είναι ευρύτερη περιοχή από το, Σιράκ, από το Ιράκ και τη Συρία. Περιλαμβάνει και την Κύπρο, το Λίβανο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη. Είναι πολύ επικίνδυνη η χρήση του όρου «Ισίλ» για την οργάνωση αυτή. Γιατί ουσιαστικά αποδίδουμε στην οργάνωση αυτή μια πολύ ευρύτερη επιρροή σε μια ευρύτερη περιοχή και ουσιαστικά μεγεθύνουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι η ίδια η τρομοκρατική οργάνωση διόρθωσε αυτό το λάθος και αντί να ονομάζεται ΙΣΙΛ, αυτό αποκλήθηκε Ισλαμικό κράτος. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον, η οργάνωση αυτή είναι μια μη συμβατική δύναμη και θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, μη συμβατική δύναμη με συμβατικό τρόπο. Θυμάστε τι έγινε με τη Μοσούλη, πώς κατέλαβαν τη Μοσούλη με 1.800 αντάρτες. Ενώ είχαμε συμβατικό Ιρακινό στρατό 55.000 στρατιωτών. Και μάλιστα έφυγε τρέχοντας ο Ιρακινός στρατός αφήνοντας και τις στολές τους ακόμη. Και οι αντάρτες ε, εισέβαλαν στη Μοσούλη και ακόμη ε, την ελέγχουν. Δεν είναι μόνο στο κομπάνι ή σε μικρές πόλεις. Ε, ελέγχουν σχεδόν το μισό Ιράκ. Το μισό Ιράκ έχει πέσει στα χέρια τους. Και το να λέμε να περιοριζόμαστε μόνο στο κομπάνι είναι σαν να θέλουμε να σκοτώσουμε κουνούπι. Ενώ ουσιαστικά πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Η πρόθεσή μας λοιπόν είναι να, ε, να εξοντώσουμε αυτή την οργάνωση για να μην έχουμε διάφορα κουνούπια αριστερά και δεξιά. Μια οργάνωση που τρομοκρατεί και απειλεί όχι μόνο την Τουρκία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο ολόκληρο. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για μας και ιδιαίτερα στο κομπάνι όπου απειλήθηκε ο κόσμος και ήθελε να διαφύγει από την πόλη για να σώσει τη ζωή του. Ανοίξαμε λοιπόν τα σύνορά μας και την πρώτη μέρα 100.000 ε, και κάτι και από το κομπάνι 138.000 συγκεκριμένα έφυγε από το κομπάνι και ήρθε στην Τουρκία. Είναι πολύ περισσότεροι οι πρόσφυγες αυτοί από όσου έλαβε η Ευρώπη από τη Συρία. Τώρα έχουμε 200.000 ε, κατοίκου πρόσφυγε από το κομπάνι στη Συρία. Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να διορθώσουμε τις εικόνες που δημιουργούμε. Γιατί μερικές φορές ε, κοιτάμε λάθος στιγμιότυπα, λάθος εικόνες. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ελέγξαμε στα σύνορα όταν έτρεχε ο καθένας για να σώσει τη ζωή του. Δεν ε, φροντίσαμε να μάθουμε αν είναι τρομοκράτη ή όχι. Ανοίξαμε απλώ τα σύνορα και ο κόσμος μπήκε στην Τουρκία και τώρα βρίσκεται στην Τουρκία. Μπορεί να είναι και... Ε, μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι απλοί άνθρωποι, να είναι μέλη του ΠΚΚ, αλλά οι άνθρωποι αυτοί θέλαν να σώσουν τη ζωή τους και ανοίξαμε τα σύνορα. Ανοίξαμε τα σύνορά μας και προς Σύριους πρόσφυγες που προσπάθησαν να διαφύγουν από βομβαρδισμούς, από δολοφονίες ε, από τη Συρία και έχουμε τώρα 1,5 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία. Μερικοί βρίσκονται σε καταβλισμούς ε, προσφυγικούς, άλλοι έχουν περάσει τα σύνορα γιατί είχαν οικογένεια, είχαν και κάποια χρήματα και προτίμησαν να μην παραμείνουν στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Ταξίδεψαν στο εσωτερικό της Τουρκίας, μερικοί πήγαν στην Άγκυρα, άλλοι στη Ισταμπούλ και μέχρι στιγμής ε, ξοδέψαμε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουμε καλύτερη ζωή στους ε, πρόσφυγες αυτές. Και δεν τους χαρακτηρίζουμε πρόσφυγες, αλλά φιλοξενούμενους μας, καλεσμένους μας. Ε, και ελάχιστες είναι οι, ε, οι συνεισφορές που πήραμε από ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, γιατί θεωρούμε ότι είναι γείτονές μας ε, οι άνθρωποι αυτοί και θέλουμε να βελτιωθεί η ζωή τους και να ρυθμιστεί η κατάσταση. Το ίδιο είχαμε και το 1998 όταν Κούρδοι Ιρακινοί, όταν χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα ει βάρο των Κούρδων Ιρακινών από το καθεστώ του Σαντάμ, 500.000 Ιρακινοί ήρθαν στην Τουρκία, έμειναν ένα χρόνο και μετά επέστρεψαν στο Ιράκ. Ανοίξαμε τα σύνορά μα και προς όσου έφυγαν από τη Βουλγαρία, οι 320.000 από του κυνηγούσε ο Ζήφκο, Ζήφκοφ. Μερικοί επέστρεψαν όταν ε, εξομαλήθηκε η κατάσταση, άλλοι παρέμειναν στην Τουρκία. Φέτος εορτάσαμε την 120η επέτειο των ε, Εβραίων Σεφαρδιτών που ήρθαν στην τουρκική επικράτεια και έκτοτε διαβιούμε ε, ειρηνικά. Αυτή, αυτό είναι το στυλ μας, αυτό είναι ο τρόπος μας. Ανοίγουμε τα σύνορά μας και θεωρούμε ότι είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο. Δεν μπορούμε όταν είναι ένα σεισμό να λέμε κάντε, να αφήσουμε τα θύματα στη μοίρα του. Αντιμετωπίζουμε και θεομηνίε. Αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν θεομηνίε και καταστροφέ από σεισμού. Τώρα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και θέλουμε να το λύσουμε. Και πιστεύω ότι ο μόνο τρόπο για να το λύσουμε είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μη συμβατική οργάνωση με μη συμβατικό τρόπο. Αν χρησιμοποιήσουμε συμβατικέ δυνάμει, δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν ε, το Ισλαμικό κράτος. Και αν δεν ε, δημιουργήσουμε ένα συνασπισμό δεν θα τα καταφέρουμε. Στο συνασπισμό χρειαζόμαστε τις Ηνωμένε Πολιτείες, χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε έτσι με έναν ευρύτερο συνασπισμό ίσως θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και συμβατικές δυνάμεις. Ελλώ, κανείς δεν θέλει να στείλει στρατιώτες και όλοι κοιτάνε την Τουρκία και κατηγορούν την ε, Τουρκία που δεν έστειλε στρατό. Δεν πρόκειται να στείλουμε τουρκικά στρατεύματα σε άλλες χώρες. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας και γι' αυτό είπαμε ας το οργανώσουμε από κοινού. Θέλουμε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή απόφαση του ΝΑΤΟ. Αλλιώς η πρότασή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε μη συμβατικές δυνάμεις που ήδη βρίσκονται στη Συρία, να διαχωρίσουμε τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης Χεσμπολά, Αλκάιντα, Ίσης και άνθρωποι που είναι ε, εκπαιδευμένοι με μη ε, συμβατικό τρόπο να χτυπήσουν αυτή την μη συμβατική οργάνωση, να τους συγκεντρώσουμε όλους, ε, να τους εξοπλίσουμε και αυτές τις μη συμβατικές δυνάμεις να στείλουμε να καταπολεμήσουν το ISIS και να λύσουμε το πρόβλημα ISIS άπαξ και διαπαντός. Αυτή είναι η πρότασή μας και ζητήσαμε ε, μία ζώνη απαγόρευσης ε, πτήσεων, no-fly zone. Και αφού θα ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και απαλλαγούμε από το ISIS, να δημιουργήσουμε μία ζώνη ασφαλείας, όχι bumper zone, ώστε μερικοί πρόσφυγες να μπορέσουν να επιστρέψουν ε, στις αιστείες τους, να επαναπατριστούν, να έχουν μια καλύτερη ζωή και να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτή είναι η πρόταση της Τουρκίας και δεν έχω ακούσει καμία αντιπρόταση. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος έχει καλύτερη απάντηση, άλλη απάντηση για αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα. Θα πρέπει όμως από κοινού να κάτσουμε και να το σκεφτούμε. Και το να στείλουμε Κούρδους αντάρτες στο κομπάνι, αυτό είναι θρύλος. Ποιοι είναι αυτοί οι Κούρδοι αντάρτες. Κανείς δεν το ξέρει. Αυτό είναι φήμε. θρύλοι. Έχουμε επαφές με το PYD, με τον Μπαρζάνη. Δεν υπάρχουν αντάρτε για να στείλουν. 55 αντάρτε ήρθαν από το κομπάνι στην Τουρκία. Ας μην μιλούμε λοιπόν με θρύλους και φανταστικά εικονικά στοιχεία, να μιλούμε με βάση την πραγματικότητα. Το θέμα το κυπριακό. Το κυπριακό πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό για μας. Και οι σχέσεις μας είναι παλιές. Εδώ και 50 χρόνια έχουμε σχέσεις και αυτό δείχνει πόσο επίμονοι, πόσο αποφασισμένοι και πόσο ανεκτικοί είμαστε. Και συνεχίζουμε αυτή τη σχέση εδώ και 50 χρόνια. Και το πρόβλημα το κυπριακό το έχουμε εδώ και 50 χρόνια. Από την τουρκική σκοπιά θέλουμε να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Και η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί από πλευρά τη. Και νομίζω ότι έχουμε μια νέα κατάσταση και νέα πλεονεκτήματα στο νησί. Καταρχήν έχουμε, ε, έχουμε βρει στον Νότο νέους φυσικούς πόρους και θα είναι ιδεώδης αυτή η κατάσταση αν όντω ε, υπάρχουν αυτοί οι πόροι και μπορούν να αξιοποιηθούν για το καλό του νησιού. Και αυτό θα είναι ένας πλούτος όχι μόνο για το νότιο τμήμα του νησιού αλλά για το σύνολο του νησιού. νησιού. Και δεν νομίζω ότι κανένας έχει αντιρρήσεις. Επίσης ε, παρέχουμε πόσιμο είδωρ στο νησί διπλάσια ποσότητα από αυτή που χρειάζεται και το βόρειο και το νότιο τμήμα θα λάβει μέχρι τα τέλη του έτους. Και φυσικά υπάρχουν κάποιες πολύ θετικέ κινήσεις. Το Φεβρουάριο οι δύο ηγέτες συνυπέγραψαν μία διακήρυξη και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Έχουμε εδώ δύο την, την λύση στο πρόβλημα και το πώς επηρεάζει το Κυπριακό της ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για να επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα ε, να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για το άνοιγμα κεφαλαίων στι διαπραγματεύσει μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για 8 χρόνια δεν καταφέραμε να, να ανοίξουμε 14 κεφάλαια επειδή κάποια στοιχεία του κυπριακού προβλήματος ε, χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμα κεφαλαίων. Εμείς θα συνεχίσουμε την στάση μας και περιμένουμε από τους Ελληνοκυπρίους φίλους και από τους Έλληνες φίλους και από τους Ευρωπαίους φίλους να δημιουργήσουν μια πιο γενική εικόνα και να δουν τα πλεονεκτήματα της κατάστασης αυτής και να συνεργαστούμε για να επιλύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Και είπα αυτή τη σκοπιά συνεχίζουμε και την ευρωπαϊκή πορεία. κάνουμε σύντομο διάλειμμα για σας. Θα είμαστε αλληλέγγυο στα δυνατόν περισσότερο. Δεν ε, είχα υπόψη ότι θα ξεπεράσουμε τόσο πολύ τα όρια του χρόνου. Είχαν προβλεφθεί 45 λεπτά για, την, ε, για αυτό το διάλογο. Ε, τελικά θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν σε πάρτε το λόγο για ένα λεπτό και μετά ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους για την κοινή συζήτηση που θα ακολουθήσει να ακούσουμε τώρα τους υπόλοιπους συναδέλφους για τα επόμενα λεπτά. Κυρία Αλιομαρή, ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι ποτέ εύκολο να προσέχετε κανεί ενώπιον μια επιτροπή σαν τη δική μα. Αλλά ήθελα να σα θέσω μια ερώτηση. Βάσει των προηγούμενων υπουργικών μου ιδιωτήτων, είχα πολύ ενδιαφέρουσε συνομιλίε με τον Τούρκο Υπουργό. Και τη στιγμή που συζητούσαμε τι σχέσει μα αυτέ, έτυχε να μου πει ότι θεωρεί πολύ απαραίτητο να έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία για να επιτευχθεί πρόοδος σε πολλά επιμέρους θέματα, αλλά επίσης στον ίδιο βαθμό από, μια μεγάλη, από ένα μεγάλο αριθμό προσώπων, πλειοψηφία μάλιστα στην Τουρκία, δεν είναι επιθυμητό η Τουρκία να έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η θέση που εκφράστηκε πριν από κάποιους μήνες ισχύει ακόμη. Ευχαριστούμε ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο των δυσχεριών που αντιμετωπίζει η διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία, με δυσκολίες που προκύπτουν όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα σας αναζήτησε μια διαφορετική ε, θέση στα γεωπολιτικά. Νομίζω ότι το πείραμα με την Αραβική Άνοιξη πριν από πολύ λίγα χρόνια δεν πέτυχε ιδιαίτερα. Τώρα βλέπουμε μια αλλαγή πορείας από την Τουρκία και προς την Ευρώπη και προς το περιφερειακό τοπίο. Αλλά υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά συγκεκριμένα στοιχεία. Φαίνεται πολύ ε, απρόθυμη Τουρκία να καταπολεμήσει τη, το ΙΖΙΣ. Αυτά που έγιναν ε, προημερών ε, με τα μέλη του ΠΚΚ είναι πραγματικά πολύ σοβαρά. Ελπίζω αυτή η διελκυστίνδα λοιπόν ε, εξουσία στην Τουρκία να επιληθεί κάποια στιγμή, αλλά έχω και μια σειρά από Τι συνέπεια υπάρχει στην ευρωπαϊκή σας θεώρηση από τη μια και από την άλλη την τάση που εφαρμόζεται στην πολιτική σας σκηνή φαίνεται να γίνεται ένας πρωταγωνιστής στις, ε, στα πολιτικά πράγματα της γεωγραφικής σας ζώνης, ε, λύοντας και δένοντας συμμαχίες. για το κουρδικό γνωρίζω τις θέσεις σας. Ε, ο στόχος δεν είναι η ανεξαρτησία, αλλά δεν είναι και καλό να χρησιμοποιείτε σημερινή συγκυρία για να περάσει η τουρκική γραμμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό βαρύνει την οποιαδήποτε προοπτική σύγκληση. Ο κύριε Στάνακο, ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι παρά την ερευνητική διαδικασία που συνεχίζεται με το ε, τοπικά κάτω του κυρίου Τσαλάν, ο πρόεδρος σας επέλεξε να περιγράψει το ΙΣΙΣ και το κουρδικό ε, κόμμα YPG ε, στο ίδιο επίπεδο, Ω τρομοκράτε και οι δύο. Ερωτώ λοιπόν το εξή: Τι υποχωρήσεις έχει κάνει η Τουρκία στο ΙΣΙΣ για την απελευθέρωση των 49 ομήρων σας και η έκκληση για μια ζώνη χωρίς πτήσεις θα ισχύει και για τα αεροπλάνα της σημασίας, της συμμαχίας που δεν πράγματα προς το ίσις γιατί αυτό προφανώς θα βοηθούσε το ίσις και θα μας εμπόδιζε μας. Σε ποιον θα ίσχυε λοιπόν αυτή η απαγόρευση πτήσεων. Σε τι αφορά επίσης την προσχώρηση της ε, ε, προς της ε, Τουρκίας στην, ε, στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη Ρωσία, τους Ταρτάρους. Ε, η Ρωσία εδώ και πολλά χρόνια είχε κρατήσει κλειστά τα σύνορα στην Αρμενία στους Αρμένιους προς αλληλεγγύη στο Αζερμπαϊτζάν. Τι γίνεται λοιπόν, τι πιστεύετε για την Ουκρανία και επίσης να πω για να μιλήσω να υποστηρίξω του συναδέλφου για τα 200 μίλια ε, αποκλειστική ζώνη για την Κύπρο. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα ήταν ατυχή και αποτελεί μια παραβίαση του κοινωνικού κεκτημένου, το οποίο η Τουρκία έχει δεσμευτεί ότι θα προσυπογράψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τάνακο, κύριε Άλλη. Ένα λεπτό, αν μπορείτε. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την θέση σας. Είμαστε πεπισμένοι για την ηγεσία σας. Όπως αναφέρθηκε, η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτώντας και εξετάζοντας τα ερωτήματα που τίθεται προς την Τουρκία, δεν είναι θέματα που άπτονται των κριτηρίων. Είναι στρατηγικά ζητήματα στη γενική περιοχή σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα της περιοχής. Αυτοί θα βαλτίουν και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι εννοώ, το πρόβλημα με τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουμε επίσης το πρόβλημα αυτό. Θα ήθελα να σας συγχαρώ λοιπόν και να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλει η Τουρκία σε ό,τι αφορά το πρόβλημα των προσφύγων. Γιατί αν η Τουρκία δεν διαδραματίσει το ρόλο της, θα υπάρξει πρόβλημα στην γενικότερη Ευρώπη. Είναι το τελευταίο σύνορο. Και κλείνω, Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όλα τα φετικά βήματα που έχουν γίνει υπό τις δεσμεύσεις σας και ότι η νέα νομοθεσία της Τουρκίας προσεγγίζει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το αντίθετο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Αλή και πολύ λυπάμαι, αλλά θα πρέπει πραγματικά να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Κύριε Βερζά, για ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε. Είναι πολύ ε, εδώ αυτοί που ανησυχούμε ε, σήμερα για την κατάσταση στη Συρία. Η αντίσταση στο Κομπάνι είναι συμβολική αξίας για την ε, απαραίτητη καταπολέμηση του Νταές του Ισλαμικού κράτους δηλαδή. Μιλήσατε για μια μη συμβατική δύναμη βεβαίως, αλλά εγώ δεν θα έλεγα ότι βγήκε και από το πουθενά. Κάποιοι ε, έκαναν τους πυροσβέστες αδίκως. Εδώ όμως πρέπει να ε, εδώ πρέπει να δούμε ε, τις προσπάθειες που γίνονται. Κανείς δεν αμφισβητεί θα έπρεπε λοιπόν να μην έχουν συναισθηματική φόρτιση, γιατί υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη στο κομπάνι και εκεί πρέπει να γίνουν ε, οι απαραίτητε κινήσει. Όταν ο Ερντογάν, ο πρόεδρο σα, λέει ότι το ΠΚΚ και το ΝΤΑΕΣ, ε, το Ισλαμικό κράτο δηλαδή, είναι το ίδιο πράγμα, αυτό δεν μα ικανοποιεί ω απάντηση. Και επιτά, όπω είπε και ο κύριο Παντζέρη, μετά του μοβαρδισμούς στην ε, κουρδική περιοχή, στι κουρδικέ περιοχέ στην Τουρκία, γιατί λοιπόν δεν αφήνετε τους Κούρδους αγωνιστές να πάνε στο κομπάνι. Λέτε ότι είναι εξεκερμένοι επαναστάτες που δεν τους γνωρίζετε. Ε, κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, η, η, η διαδικασία σε συνεργασία με το ΠΚΚ πώς, πώς προχωρεί. Τα πράγματα δεν μου φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Εδώ θα θέλαμε να είστε πολύ σαφείς στην απάντησή σας για να καταλάβουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Καστάλντο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σας Υπουργέ. Θα ήθελα να επαναφέρω και το θέμα των διαπραγματεύσεων, διότι το έχουμε συζητήσει και με τον Επίτροπο Φίλε μόλις την περασμένη εβδομάδα από μια χώρα που έχει τεράστιους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με την Τουρκία, την Ιταλία, θεωρώ θετικό η Τουρκία να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Όμως, όπως είπε και ο συνάδελφος Εμπάγιας προηγουμένως, ακόμη και αν είμαστε καλοί φίλοι πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας. Οπότε πρέπει να φυγούν ε, και τα πιο ακαθόδη ζητήματα με τον Επίτροπο Φίλε. Είχαμε συζητήσει και τη δυνατότητα να γίνει πρόοδο στα κεφάλαια 23 και 24 για τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα θεμελιώδη μάλλον δικαιώματα. Γιατί στον ποινικό σα κώδικα δεν υπάρχει ένα σαφής ορισμός ε, της ε, στο εδάφιο ε, 91. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας βασικός πυλώνας του κράτος δικαίου που θα πρέπει να υπάρχει. Και επίσης τι θα γίνει με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στη χώρα και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί προσφάτως. Και κυρίω τη διεξαγωγή τη προκλητική εκστρατεία. Αναφέρομαι στο YouTube και στο Twitter. Θα πρέπει Επίσης να σχολιάσετε και την επιλογή της Τουρκίας να μην, ε, να μην παρέμβει στο κομπάνι και να μην επιτρέψει την πρόσβαση των ε, Κούρδων αγωνιστών σε αυτήν την περιοχή για να προσφέρουν ενισχύσεις. Πώς το εξηγείτε. Ευχαριστούμε συνάδελφε Καστάλντο, ο κύριος Επιτίδιος. Αλλά παρακαλώ 50 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό οι περισσότερες παρεμβάσεις γιατί πραγματικά έχουμε περβεί κατά 15 λεπτά τουλάχιστον το χρόνο. Κύριε Υπουργέ, είπατε προηγουμένως ότι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας θα επιδιώξετε να αλλάξετε την εικόνα που επικρατεί για τη χώρα σας στην Ευρώπη. Ε, θα ήθελα να παρατηρήσω όμως ότι η, Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα με πόλεμο εάν αυτή ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει σε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά της ύδατα. Επίσης αρνείστε την οντότητα μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσης της Κύπρου, της οποίας η Τουρκία κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους. Πρόσφατα ο κύριος Νταβούτογλου είπε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πληρώσει τα χρήματα τα οποία επεδίκασε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις ζημιές που προκάλεσε η εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Τέλος, ε, η Τουρκία δεν ελέγχει, παρά το γεγονός ότι λαμβάνει σχετικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σύνορά της με την Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε μέρα να σειραίνουν εκατοντάδες λαθρομετανάστες εκεί. Πώς πιστεύετε ότι αυτή η, η τακτική θα βοηθήσει την προοπτική την ευρωπαϊκή της Τουρκίας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Λένερτς και Μαυρίδης παρακαλώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Δύο σύντομε ερωτήσει έχω. Στον έγγραφο στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάτε για την ανάγκη νέου συντάγματο. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένω εδώ, αλλά φαίνεται ότι δεν προχωράει η διαδικασία στην Τουρκία. Έχει παγώσει. Τι θα κάνετε για να αναζωογονήσετε ή να ξεκινήσετε εκ νέου αυτή τη διαδικασία. Είπατε θα έχετε στενή συνεργασία και διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν αποφασίζετε νέες νομοθετικέ διατάξεις σε ό,τι αφορά τις αλλαγές για το είπα το Συμβούλιο εισαγγελών και Δικαστών που κρίθηκε αντισυνταγματικά. Πώς το βλέπετε αυτό. Γιατί οι μεταθέσεις ε, δικαστών και εισαγγελέων ήδη έγιναν. Ε, πώς θα λάβετε υπόψη στις τάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης μελλοντικές σας ε, νομοθετικές διατάξεις. Ο κ. Μαυρίδης. Είμαι σύντομος. Άκουσα τη φράση που είπατε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πραγματικότητες και όχι θρύλους. Δύο πραγματικότητες εδώ. Το 2005 είχαμε διαπραγματευτικό πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Το πλαίσιο αυτό προέβλεπε συγκεκριμένες ε, υποχρεώσεις. Έχουν περάσει εννέα χρόνια και δεν έχουν τηρηθεί αυτές οι υποχρεώσεις. Ποια είναι τα σχόλιά σας. Δεύτερον, μια άλλη πραγματικότητα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος, ο Λίβανος, ε, το Ισραήλ και η Αίγυπτος συμφώνησαν ε, για καταμερισμό των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με βάση τον, το δίκαιο της θάλασσας που αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού και Θα σεβαστείτε τα δικαιώματα των χωρών αυτών που στηρίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία ή θα το καταπατήσετε. Τα πράγματα είναι απλούστατα. Θέλουμε και εμείς πραγματικότητες. Ο κύριος Μποργέτσιο. Υπουργέ, όπως ξέρετε καλά, Ιζιλ ή Ιζις, όπως και αν το πούμε, δεν είναι μια απειλή μόνο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής του παλιού Λεβάντε. Αλλά είναι για ε, όλη την, ε, για το δυτικό χριστιανισμό. Με μια μαύρη σημαία η οποία θα νεμίζει υποθετικά κάποια στιγμή στο μέλλον και στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης στο Βατικανό. Ε, εδώ λοιπόν δεν βοηθάτε τους ε, Κούρδους στο κομπάνι. Ντροπή σας Τουρκία, ντροπή σας να ντρέπεστε. Ευχαριστούμε κύριε Μποργέτσιο, αλλά ας προσπαθήσουμε να είμαστε ευγενεί και κόσμοι εδώ. Ο κύριος Παπαδάκης. Ε, πολύ θα χαιρόμουν να είχαμε μια νέα Τουρκία. Αντίθετα, εντείνεται η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας με την παρουσία πολεμικών πλοίων τη στιγμή αυτή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και καταπατάτε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η μη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς μας αποδεικνύει ότι δεν θέλετε ουσιαστικά να μπείτε στην Τουρκία. Κάντε κάτι ούτως ώστε να είμαστε στην ίδια μεριά, να μπει η Τουρκία με το σεβασμό στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τάσεις σας επιδεικνύεται ότι θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί στις δικές σας πολιτικές πρακτικές. Και κάτι τελευταίο για το ISIS. Αν θέλατε να σκοτώσετε τα κουνούπια θα μπορούσατε να ψεγάσετε. Okay. Thank you. Thank you very Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδάκη και η συζήτηση αυτή λοιπόν ολοκληρώθηκε. Θα ζητήσω από τον Υπουργό τώρα να κάνει το αδύνατον, να προσπαθήσει να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις σε 5 έως 7 λεπτά και φαντάζομαι ότι το ηθικό δίδαγμα ε, είναι ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να προβλέψουμε πολύ πιο πολύ χρόνο. Ζητώ συγγνώμη και πάλι στους συναδέλφους της ΛΥΜΠΕ που είναι εδώ. Σας παρακαλώ, λοιπόν, έχετε το λόγο για καταλεκτικά σχόλια σας. Ε, Ευχαριστώ. Μα ήταν ερωτήσει 20 ε, λεπτών. Πώ θα τι απαντήσω σε 5 λεπτά. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Καταρχά, δεν θέλω να μπω στην ίδια παγίδα και να χρησιμοποιήσω το ίδιο ύφο στην επιτροπή αυτή και να απαντήσω με τα ίδια λόγια. Καταρχά, το ΠΚΚ και το ISIS, οι σχέσει του. Το ΠΚΚ είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει ανακηρυχθεί από τον ΝΑΤΟ, από τη ΣΥΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τρομοκρατική οργάνωση. Ο κύριος Τάνοκ θα έχει ξεχάσει ίσως τι έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο για να αντιμετωπίσει το Ιρλανδικό πρόβλημα. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Η τρομοκρατική οργάνωση και το πολιτικό κόμμα α, κλήθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιληθεί το πρόβλημα. Και όταν ε, είχαμε τι βόμβε στο Λονδίνο, το ίδιο συνεχίσατε να κάνετε. Τι κάνουμε λοιπόν, το ΠΚΚ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Μαζί με το πολιτικό του σκέλος στο Κοινοβούλιο γίνονται διαπραγματεύσει και η ειρηνευτική διαδικασία συνεχίζεται. Θα πρέπει να δείτε στην έκθεση προόδου όπου ε, τονίζονται οι δυτικέ εξελίξει και ανεξαρτήτως πώ θα συνεχίσουμε τις ε, διαδικασίες αυτές, την ερευνητική αυτή διαδικασία, γιατί είναι προ όφελο των ε, πολιτών της Τουρκίας κουρδικής καταγωγής, υπέρ του Βόρειου Ουρα, Ιράκ, της περιφέρειας, της περιοχής και για το μέλλον της Τουρκίας άλλωστε. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Αυτό που αναφέρατε για την τουρκική υποστήριξη, κυρία μου, για την ε, ευρωπαϊκή διαδικασία. Στην Τουρκία σε καμία χρονική περίοδο ε, οι πολέμοι της προσχώρησης στην Ένωση δεν έφτασαν πάνω το 10%. Αυτό που άλλαξε είναι η αναποφάσιστη. Έχουμε 5-55% υποστήριξη πλέον. Αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι συνεχίζει να κινείται το όχημα και έχει φύγει, αν θέλετε, το πλοίο από το λιμάνι, αυτό το ποσοστό των αποφάσεων θα μειωθεί για τις πολλαπλές ε, λοιπές ερωτήσεις σας. Πολύ θα ήθελα να εξηγήσω. Αν μου δώσετε χρόνο, ευχαρίστως να το κάνω. Σε πέντε λεπτά όμως μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω ουσιαστικά. Για το νέο σύνταγμα, για παράδειγμα, το οποίο έθιξε ο κύριος Λέναρτς, σημειώθηκε πρόοδος. Δεν το πετύχαμε, αλλά στις επόμενες εκλογές, αν το κόμμα μας λάβει την απαραίτητη πλειοψηφία προκειμένου να κάνει δημοψήφισμα. Δεν έχουμε τώρα αυτή την πλειοψηφία αυτή. Θα εργαστούμε για ένα νέο σύνταγμα. Ετέθησε ένα ερώτημα επίσης για την Τουρκία. Γιατί ε, έκανε η Τουρκία για να πετύχει τη συμφωνία της Μουσούλης. Έχουμε 59 άτομα που είναι στα χέρια της ίσης και εργάζονται για το τουρκικό συμβούλιο. 49, συγγνώμη. Αν είχε καλές σχέσεις θα τους κρατούσαν. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που κάνει πρωτίστως μια χώρα να έχει ομήρους είναι να σώσει τους ομήρους. Και κάθε χώρα λοιπόν κάνει τέτοιου είδους ε, συμφωνίες. Τι κάναμε για να σώσουμε 49 ζωές. Είναι μια απόρριτη συμφωνία αυτή. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Και το νομίζω Βασίλη τα έχει κάνει και πολλέ άλλε χώρε τα έχουν κάνει. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να μας απαιτήσετε ευθύνε γι' αυτό. Τώρα, για τις ε, κυρώσεις στη Ρωσία. Είμαστε απολύτως αντέθετοι σε οποιαδήποτε κατοχή εδάφους άλλης χώρας. Ανοιχτά δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία τονίζουμε ότι ε, υποστηρίζουμε την πολιτική σταθερότητα και την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Αλλά από την άλλη δεν πιστεύω προσωπικά ότι οι κυρώσεις είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δεν είχαν ε, ούτε στη Λιβύη, ούτε στη Συρία, ούτε στο Ιράκ αποτέλεσμα, ούτε στο Ιράν αποτέλεσμα οι κυρώσεις. Άρα αν επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Και πολλές χώρες ε, έχουν συμφέροντα και οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν ε, θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με τι κυρώσει αυτέ, όταν οι αποφάσει αυτέ ελήφθησαν χωρί την παρουσία μα. Μα παρουσιάστηκαν. Απλά για να τι εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι για να κρατήσουμε τη Ρωσία στο παιχνίδι δεν πρέπει να εφαρμόσουμε κυρώσεις αλλά να αυξήσουμε τα κίνητρα. Να προσέξουμε γιατί παίζουν σκάκι καλύτερα από κάθε άλλο οι Ρώσοι ξέρετε. Καλύτερα από κάθε άλλη χώρα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Τώρα λόγω των κυρώσεων αυτό το σκάκι θα το παίξουν για να μας αναγκάσουμε να παίξουμε ρωσική λουλέτα. Επιλύ... προσπαθώντας να επιλύσουμε λοιπόν το πρόβλημα της Συρίας, το πρόβλημα του Ίσης, δεν θα πρέπει παράλληλα να ξεχνάμε ποια είναι η επιρροή της Ρωσίας εκεί. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα πρέπει να πείσουμε τη Ρωσία να συμμετάσχει στην όλη ιστορία. Χρειάζομαι απόφαση του Συμβουλίου ασφαλεία του ΟΗΕ, συμμετέχει η Ρωσία, να σταματήσουμε την παράδοση όπλων στους, ε, στις αρχές της Συρίας και πάλι είναι η Ρωσία. Όπου και να κοιτάξουμε παντού είναι η Ρωσία. Αν τους βάλουμε στη γωνία η απάντηση θα είναι ότι δεν θα επιληθούν προβλήματα. Προβλήματα που εμείς θέλουμε να επιληθούν. Πόσο χρόνο έχω πρόεδρε. Δύο λεπτά. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομικό σύστημα, το σύστημα Τη δικαιοσύνη στην Τουρκία. Αυτό που έγινε την προηγούμενη Κυριακή θεωρώ ότι αποτελεί μια καλή απόδειξη για το γεγονός ότι σωστά λειτουργεί το δικαστικό σώμα. 14.000 ε, δικαστές ψήφισαν και σε ό,τι αφορά το σύστημα αυτό. Και νομίζω ότι αυτό που τελεί μια καλή απόδειξη στο ότι μπορεί να γίνει δημοκρατικά η διαδικασία αυτή είναι βασική μας ε, ανησυχία. Να υπάρχει δικαστικό σώμα αξιόπιστο, έντιμο, στο οποίο να μπορούμε να βασιστούμε. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της τριετίας, όπου αντιμετωπίσαμε δυσκολίε σε ό,τι αφορά την διαδικασία Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε πάνω από 60 πακέτα τα οποία περιείχαν στοιχεία για την ανεξαρτησία του δικουστικού σώματος. Το 2009 υπήρξε στρατηγική για την δικαστική μεταρρύθμιση. Ανανεώνεται, εφαρμόζεται προκειμένου το δικαστικό σύστημα που αποτελεί βασικό πυλώνα για την οικονομία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιαδήποτε χώρα να είναι ανεξάρτητο και δίκαιο. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση σε άλλο ένα ερώτημα. Πάνε και τα δύο λεπτά μου. Σας παρακαλώ, προσκαλέστε με και πάλι για να με ερωτήσετε ξανά πράγματα, αλλά δώστε μου λίγο παραπάνω χρόνο όταν μου θέλετε τα ερωτήματα. Με μεγάλη μου χαρά. Μη μου πείτε, μην ναι, πείτε μεταξύ σας όταν φύγω ότι έφυγε και δεν απάντησε στις ερωτήσεις μου. Δεν μου δίνει ο πρόεδρος χρόνο. Αυτός φταίει. Μάλιστα. Αναλαμβάνω την ευθύνη, λέει ο πρόεδρος. Γιατί τα θέματα τα οποία δεν απαντήθηκαν και τα οποία ετήχθησαν σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Υπουργέ, όλοι κατανοούμε νομίζω ότι οι τουρκικέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ εξ ορισμού και το ότι οι περιφερειακέ σχέσει τις περιπλέκουν περαιτέρω. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μελλοντική ευκαιρία και θα σα προσκαλέσουμε εκ νέου στην Επιτροπή μα για να συζητήσουμε, ζητώ και πάλι συγγνώμη στους συναδέλφου τη ΛΥΜΠΕ, για την καθυστέρηση διάλειμμα ενό λεπτού και συνεχίζουμε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 Ευχαριστούμε πολύ. Ας προσπαθήσουμε να ησυχάσουμε στην ε, αίθουσα. Όσοι δεν θα μείνουν για αυτό το μέρο τη ε, συνεδρίασης, παρακαλώ ε, φύγετε ήσυχα από την αίθουσα. Παρακαλώ να καλωσορίσω επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τον κύριο Ζαν Λαμπόρντ από τον ΟΗΕ. Είναι εκδοτικός διευθυντής του τη Εκτελεστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση τη Τρομοκρατία. Είναι μεγάλη μα χαρά να σα υποδεχόμαστε εδώ για την κοινή συνεδρίαση ΛΥΜΠΕ και ΑΘΕΤ και να καλωσορίσω και τον πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, τον κύριο Κλοντ Μωράη και τα μέλη της Επιτροπής του για την υπομονή τους μόλις τώρα. Κύριε Λαμπόρντ, χθε είχατε συναντήσεις και με εκπροσώπους των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων και νομίζω ότι οι εκπρόσωποι και των δύο επιτροπών μας έχουν μεγάλη περιέργεια να ακούσουν τι έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των, της και των εσωτερικών αλλά και των εξωτερικών μας σχέσεων για την, ε, θέσπιση μέτρων κατά της θερμοκρατίας την Δευτέρα και την Τρίτη. Ε, οι εισαγγελείς ε, του Βελγίου, της Γαλλίας και της Ισπανίας συναντήθηκαν στην Κόρτοβα για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους. Δεν θα είναι έκπληξη για τους συναδέλφους της ΛΥΜΠΕ ε, που η δημιουργία σχέσεων με τις χώρες της άμεσης γειτονιά μας είναι πρώτη προτεραιότητα και για την καταπολέμηση του ΆΙΖΙΣ και για τον εξωτερικό μας την εξωτερική μας άμυνα. Ελπίζω λοιπόν υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στη Συρία και το Ιράκ να έχουμε σήμερα χρήσιμες πληροφορίες. Να πούμε ότι οι τρομοκράτες συνήθως ξεκινούν από την εικασία ότι ε, μάχονται ένα δίκαιο πόλεμο, ότι έχουν το δίκαιο με το μέρος τους και ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα περισσότερες χώρες όμως ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ασχολούνται με τρομοκρατικές ομάδες που μόλις έχουν δράσει, σκοπεύουν να δράσουν, ε, υπάρχει απειλή ότι θα δράσουν, αλλά πρέπει να είμαστε και περισσότερο προσεκτικοί με το σκέλος της πρόληψης. Γι' αυτό λοιπόν οι μέσα σα θα είναι πολύ χρήσιμες για τη σημερινή μας συζήτηση και καλό θα να σχολιάσουμε όλους τους μηχανισμούς που διαθέτουμε από τις ηρεμιστικές υπηρεσίες μέχρι τα κλασικά μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επίσης κάτι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προστασία των συνόρων μας. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή και για αυτούς που εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να γνωρίζουμε πού κατευθύνονται. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, λίγα λόγια εισαγωγικά ήταν αυτά. Κύριε Μωράης, έχετε και εσείς το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Πλέγκοβιτς. Ε, είναι νομίζω πολύ χρήσιμο να έχουμε μια κοινή συνεδρίαση της ΑΦΕΤ ε, και της Επιτροπής Ελευθεριών του Πολίτη για τα θέματα αυτά. Καλωσορίζω τον Ζαν Πολαμπόρντ εκ μέρους των ε, μελών της δικής μου επιτροπής, της ΛΥΜΠΕ, είναι θέμα ιδιαίτερης σημασίας αυτό για μας ε, και η συνεργασία μας με την ΑΦΕΤ βεβαίως, αλλά εδώ έχουμε κέρι ε, αρμοδιότητα επί των ζητημάτων αυτών. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι σαφώς εθνική αρμοδιότητα. Θα μας το πει και ο Ζαν Λαμπόλα φαντάζομαι, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη έχουν ε, και προβλέπουν νομοθετικές ε, κινήσεις ε, και νόμους για το θέμα αυτό, αλλά και η κοινή μας στρατηγική είναι ένα θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο και σημαντικό. Για τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ είναι μια σοβαρότατη αρμοδιότητα που έχουμε αναλάβει και γι' αυτό θέλουμε την ανταλλαγή απόψεων που οργανώθηκε σήμερα. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, διότι και το Μητρό Επιβατών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών όλα τα θέματα προστασίας του ιδιωτικού βίου και ασφάλειας το τι θα σημάνει μια τέτοια στρατηγική κοινή με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις Ε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες του θέματος. Έχουμε λοιπόν και εμείς αρμοδιότητες εδώ και ε, αναμένουμε με ιδιαίτερη προσοχή τη συζήτηση αυτή. Δεν θέλουμε να είμαστε ε, αρνητικοί καθόλου στην τοποθέτησή μα. Είναι ένα θέμα βεβαίως που προκαλεί την προσοχή μας και μα κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι ένα θέμα για όλα τα μέλη της Επιτροπής μας που έχει αυτό το χαρακτήρα, αλλά είναι σημαντικό και για την εσωτερική πολιτική ασφάλειας που θα έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείτε ότι θα συμβεί αυτό και από τι ερωτήσει που θα τεθούν. Σα ευχαριστώ πάντω για την παρουσία σα σήμερα και, για την... και ευχαριστώ και του συναδέλφου τη Επιτροπή ΑΦΕΤ για την ε, καλή συνεργασία που έχουμε. Κύριε Λαμπόρντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Πρόεδροι μάλλον, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την σημερινή μου παρουσία και τη τιμή αυτή δυστυχώς ε, την αντλάω από το γεγονός ότι θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη απειλή. Και στις εισαγωγές σας το επισημάνατε και γι' αυτό βρίσκεστε και οι δύο παρόντες. Το θέμα δεν είναι μόνο εξωτερικό. Ούτε είναι μόνο εσωτερικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα αυτό έχει και εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές και η απειλή είναι πραγματικά τεράστια. Δεν θα αναφέρω εδώ αριθμητικά στοιχεία, ούτε χρειάζεται να επιμείνουμε στις διαστάσεις της απειλής, γιατί είναι γνωστές αυτές σε όλους. Έχουμε πάνω από 10.000 ε, μαχητές, τρομοκράτες, ε, ξένοι τρομοκράτες, το τονίζω αυτό, μαχητές ε, έχουν πάει στη Συρία και το Ιράκ. και βέβαια ακριβή στοιχεία δεν έχουμε, αλλά υπολογίζουμε ότι έχουμε 2 με 3 χιλιάδες ε, ξένους τρομοκράτες μαχητές ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όμως ε, η μόνη ή η πιο σημαντική μερίδα τους. Η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο τμήμα των ξένων μαχητών προέρχονται από τις χώρες του Μαγκρέπη της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι τόσο από την Ευρώπη αυτοί οι ξένοι μαχητές ή από την Ομοσπονδία της Ρωσίας, από την Κίνα επίσης προέρχονται ξένοι μαχητές. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι αποκλειστικό πρόβλημα της Ευρώπης, αλλά είναι και ευρωπαϊκό το πρόβλημα, γιατί πολύ εύστοχα επισημάνεται ότι υπάρχουν ζητήματα διαχείρισης των συνόρων, που είναι κέρια σημασίας και για σας και φυσικά υπάρχουν και θέματα που άπτονται αυτής της ισορροπίας που ουσιαστικά ισοδυναμεί με τετραγωνισμό του κύκλου. Πώς θα βρούμε την ισορροπία μεταξύ των απαραίτητων μέτρων και του σεβασμού των δημοσίων των πολιτικών ελευθεριών. Και δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών ελευθεριών, είναι θέμα σεβασμού των ιδρυτικών μας αρχών και αξιών και όχι μόνο των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των μελών του ΟΗΕ γιατί έχουμε τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών έχουμε τη χάρτα των ε, πολιτικών ε, δικαιωμάτων που επίσης είναι η οικουμενική χάρτα και έχουμε και την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλες οι χώρες ε, που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν τον ίδιο, την ίδια αντίληψη για τη σπουδαιότητα που έχει η ανέβρεση αυτής της ισορροπίας. Θα μπορούσα και εδώ να σταματήσω αν δεν ήμουν υποχρεωμένος να αναφερθώ και στα επιμέρους ζητήματα. Όπως είπατε, είμαι ο εκτελεστικός διευθυντής της Εκτελεστικής Επιτροπής. Βέβαια, λίγο βάρβαρα ακούγονται όλα αυτά, όπως όλα τα αρχικά των διεθνών οργανισμών, της Εκτελεστικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και έχω άμεση σχέση και με την αντίστοιχη επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας και ουσιαστικά αναφέρομαι στην ε, ε, Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είχαμε το ψήφισμα 2178 μετά τη Σύνοδο Κορυφής που έγινε πριν από τρεις εβδομάδες στη Νέα Υόρκη και εκεί οι 15 ε, χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κατέληξαν σε ένα κοινό ψήφισμα που αφορά το κεφάλαιο 7 και σας ενδιαφέρει, πρόκειται για ένα δεσμευτικό ψήφισμα, δεσμευτικό, binding, τουλάχιστον για το διατακτικό του σκέλος και επίσης το ψήφισμα αυτό περιλαμβάνει κάποια πολύ σημαντικά σημεία και για σας. Υποχρεώνει τα κράτη-μέλη καταρχήν επισημαίνει πρώτα απ' όλα ότι όλοι είμαστε ενωμένοι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο των ε, ξένων τρομοκρατών μαχητών. Αλλά δεν θα πρέπει να απομονώσουμε ε, ή να εξατομικεύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δίνουμε ε, γενικότερη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Και είχαμε το πρώτο ψήφισμα του Συμβουλίου το 1373, το πρώτο ψήφισμα για την τρομοκρατία και θα πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο θέματα. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίζουμε. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε πλήρως το θέμα των ξένων τρομοκρατών μαχητών από τις ε, πρακτικές που έχουμε και τις ήδη τρέχουσες εργασίες κατά της τρομοκρατίας. Φυσικά έχουμε το εύρος αυτού του φαινομένου και τις διαστάσεις του, το φαινομένου των ξένων μαχητών δηλαδή που μας ευνηδίασε και που αφορά την πολιτική με επίκεφαλαίο και όχι την πολιτικά και την κομματική πολιτική. Οπότε αυτή η μάχη που δίνουμε δεν είναι μόνο η μάχη κατά του Ισίλ, του υποτιθέμενου Ισλαμικού κράτους. Και λέω υποτιθέμενου γιατί μερικές φορές ερμηνεύουμε ε, κάποιους όρους, γιατί η οργάνωση αυτή έχει κάποιες δομές που μπορεί να προσωμιάζουμε τις δομές ενός κράτους, αλλά δεν θα πρέπει να δώσουμε στην οργάνωση αυτή το προνόμιο ή την τιμή και να την αποκαλούμε κράτος. Πάνω απ' όλα πρόκειται για μια οργάνωση, τρομοκρατική μάλιστα οργάνωση, μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει κάποιες διαρθρώσεις που μοιάζουν με κρατικές δομές, αλλά στην ουσία δεν είναι κράτος η οργάνωση αυτή. Ένα το κρατούμενο. Υπάρχουν όμως και άλλες ε, οργανώσεις. Η Μπόκο Χαράμ στην Ιγερία, Άγνη, δεν θα τις αναφέρω όλες. Η καταπολέμηση λοιπόν της τρομοκρατίας είναι ένας ευρύτερος αγώνας που καλούμαστε να διενεργήσουμε. Τώρα, πώς μπορώ να σας βοηθήσω και πώς ε, να προσφέρω εδώ μια προστιθέμενη αξία στην όλη συζήτηση. Και για να οικονομήσω και την ομίγυρη θα, θα συνεχίσω ίσως και στα αγγλικά κάποια στιγμή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η εκτελεστική επιτροπή συστήθηκε το 2005 που στόχο έχει την, ε, επι, την ε, επιτήρηση των τρομοκρατικών μέτρων, της παροχής τεχνογνωσίας, ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών και στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους. Και γι' αυτό έχουμε στενή συνεργασία με την Interpol, την Europol, την Εξωτερική Υπηρεσία ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με τους συντονιστές και δεν έχουμε απλώς συνεργασία, και μια, βρισκό, μια και είμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλεία και θέλουμε να εκτιμήσουμε τις ικανότητε των κρατών μελών και να προσφέρουμε και τεχνική αρρωγή, έχουμε επισκέψεις, πραγματοποιούμε επισκέψεις στι διάφορες χώρες. Πήγαμε πρόσφατα στην Μάλτα, την επόμενο μήνα θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στη Γαλλία. Δηλαδή, όλα όσα κάνουμε δεν είναι να ε, στυλιτεύσουμε τις αδυναμίες των χωρών μελών να εφαρμόσουν αντιτρομοκρατικά μέτρα ή να καταπολεμήσουν τη δρομοκρατία, τονίζουμε και τις βέλτιστες πρακτικές και προσπαθούμε να μιμηθούμε ή να γενικεύσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Μέχρι στιγμής ε, έχουμε ε, επισκεφθεί πολλές χώρες μέλη και θα συνεχίσουμε το διάλογο με τις υπόλοιπες χώρες μέλη Έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 100 επισκέψεις και θα συνεχίσουμε τις επισκέψεις αυτές. Ένας τομέας πολύ ευαίσθητος και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαντάζομαι και απόδειξη είναι η παρουσία εδώ του Προέδρου της ε, Επιτροπής Πολιτικών Ελευθερίων. Πώς το λέτε, πώς το λέτε, πώς λέτε την Επιτροπή. Δεν το ξέρετε εσείς που είστε Άγγλος, εγώ τι να πω τότε που είμαι και Γάλλος. Οπότε, ό,τι συγκεντρώνουμε ε, από την αντιτροποκρατική μας εμπειρία το χρησιμοποιούμε αλλά με γνώμονα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάτι που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερος και απόδειξη η σημερινή αυτή κοινή συνεδρίαση και σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση των συνόρων και φυσικά αυτό το θέμα το λαμβάνουμε υπόψη πολύ συχνά το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρείται ότι ασχολείται μόνο με θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Και παραμελούμε πολλές φορές το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας φροντίζει ιδιαίτερως και μεριμνά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα για επιμέρους πτυχές των αντιτρομοκρατικών μέτρων. Στο πρώτο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το 1373, που ελήφθη μετά το, την 11η ε, Σεπτεμβρίου του 2001, το πρώτο αυτό ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό. Λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε όλοι όσοι συμμετέχουν σε τρομοκρατικές ενέργειες να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πρώτη αρχή. Και σε άριθμα άλλα ψηφίσματα αναφέρεται ότι τα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας θα πρέπει να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερως το ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο για τους πρόσφυγες και τα διεθνή δικαιώματα. Οπότε στις αξιολογήσεις που κάνουμε εντοπίσαμε τι γίνεται με τις ε, ανακριτικές εξουσίες και ερευνητικέ των κρατών μελών και κυρίως ό,τι αφορά την παραπομπή των ε, υπόπτων τρομοκρατίας στη δικαιοσύνη. Σε πολλές περιπτώσεις ε, έχουμε κράτη-μέλη που ε, υιοθέτησαν ειδικέ αντιτρομοκρατικές ε, νομοθεσίες, ενώ άλλε χώρες αναθεώρησαν υπάρχουσα νομοθεσία προκειμένου να διευρύνουν τις εισαγγελικές ε, ανακριτικές εξεταστικές του αρμοδιότητες. Τώρα, τι μέτρα λαμβάνονται. Έχουμε αυξανόμενη επιτήρηση με εποπτεία και ιδιαίτερες ε, ε, ε, αρμοδιότητες υπηρεσίες πληροφοριών σε πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών και διευρυμένες εξουσίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Τι λένε τώρα οι οργανισμοί και οι τροπές του ΟΗΕ για τα θέματα αυτά, για τις γενικές αυτές πρακτικές. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι περιφερειακοί μηχανισμοί έχουν τονίσει ότι η χρήση ειδικών διαδικασιών και κυρίως εκείνων που περιορίζουν την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο ε, για την υλοποίηση εύλογου στόχου και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της αναγκαιότητας, πολύ σημαντικό, της αναλογικότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Αυτό προσπαθούμε κάθε φορά να εφαρμόζουμε. Επίσης, οι ειδικέ διαδικασίες των χωρών θα πρέπει να διαχωρίζονται από τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση εθνικών εκτάκτων αναγκών που και που προβλέπουν παρέκκληση από μερικέ υποχρεώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με βάση το άρθρο 4 του Διεθνού Συμφώνου για τι Πολιτικέ Ελευθερίε και τα Πολιτικά Δικαιώματα προβλέπεται ότι έκτακτα μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο σε περίπτωση όμω εθνική εκτάκτου ανάγκη μία εκτάκτου ανάγκη που απειλεί την, τη ζωή των πολιτών και με βάση επίσημη, ε, επίσημη διακήρυξη. Και μάλιστα τα έκτακτα μέτρα υπόκειται σε αυστηρές προποθέσει, και μάλιστα δεν επιτρέπονται εξαιρέσει για ορισμένα δικαιώματα. Και τέλος, ό,τι αφορά την αναγκαιότητα των μέτρων και την αναλογικότητά τους, περιορισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει περιορισμένο χρόνο και να υπόκειται σε πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις. Αυτό λοιπόν κάνουμε, αυτή την επιτήρηση και αξιολόγηση και κάθε φορά που πραγματοποιούμε επίσκεψη επισημαίνουμε αυτά τα μέτρα και υποβάλλουμε και κάποιες συστάσεις. Συνήθως ε, συστήνουμε συστηματική αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας προκειμένου να καλυφθούν, να γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις από το, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά καλύπτουμε εδώ τις υποχρεώσεις όχι μόνο των κυβερνητικών φορέων αλλά και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα πρέπει στο διάλογο αυτό να εμπλέκουμε και την κοινωνία των πολιτών πριν θεσμοθετηθούν έκτακτα μέτρα και φυσικά να υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί και ρήτρε εκπνοής για ειδικά τέτοια μέτρα και επίση ζητούμε την δημιουργία ή την ενίσχυση του ανεξάρτητου ελέγχου και των φορέων εποπτείας και φυσικά και προβλέπουμε και τη θέσπιση ειδικευμένων προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ψήφισμα 2178 του Συμβουλίου Ασφαλεία, το ψήφισμα αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δεσμευτικό και αφορά το μηχανισμό των ξένων μαχητών. Το ψήφισμα αυτό του ΙΕ έχει συμπεριλάβει και τα συγκεκριμένα στοιχεία που σας προανέφερα στο, ε, στο διατακτικό του, δηλαδή το στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι άλλο που τονίστηκε και αναφέρεται και στο ψήφισμα αφορά τα αντιτρομοκρατικά μέτρα. Ή το θέμα της, του διαδικτύου Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τον φανατισμό και τον εξτρεμισμό, τον βίο, με συγκεκριμένη ρητορική. Γι' αυτό και καλέσαμε στη Νέα Υόρκη το, τους Υπουργούς Θρησκευτικών Υποθέσεων του Μαρόκου, της Γουινέας, του Μαλή, της Μαυριτανίας και της ακτής του Ελεφαντοστού. Τους προσκαλέσαμε στην Νέα Υόρκη και εκείνοι που είναι μουσουλμάνοι δήλωσαν και όχι εμείς ότι η Ισλαμική θρησκεία είναι μια ειρηνική, φιλειρηνική θρησκεία. Και μάλιστα έχουν προγράμματα που εκπαιδεύουν τους ημάμιδες πριν αναλάβουν συγκεκριμένες θέσεις σε χώρες. Κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης έχουν εκπαιδεύσει ημάμιδες στο Μαλί και σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία που εκπορέθηκε από τις χώρες αυτές για να καταπολεμηθεί ο φανατικός εξτρεμισμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο βίος εξτρεμισμός πρέπει να καταπολεμηθεί. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την υπομονή σας και την παράταση του χρόνου που μου δώσατε και ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Διευθυντά. Ήρθατε από τη Νέα Υόρκη και μας περιμένατε και 30 λεπτά. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αλλά δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από τις χρονοθερίδες που προβλέπονται. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσίασή σας, για όλες αυτές τις εξηγήσει, για το ψήφισμα 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας που είναι άκρο σημαντικό στο σημερινό πλαίσιο για την καταπολέμηση τη δημοκρατία. Εάν λοιπόν μου επιτρέπετε κύριε Μωράης να δώσω το λόγο απευθείας στη συνάδελφο κυρία Γκόμες από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Λαμπόρντ, να ρωτήσω. Τονίζετε την ανάγκη να υπάρχει μια σφαιρική, μια συνολική προσέγγιση όχι μόνο της εσωτερικής ασφάλειας πια, αλλά να είμαστε ολιστικοί στην προσέγγιση μας. Δηλαδή, οι μέρημνες της εξωτερικής πολιτικής να συνάδουν και να συνδυάζονται με την εσωτερική και να προλαμβάνουμε αλλά και να επιλύουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Τώρα, μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με του με τους ξένους μαχητές ε, στην περίπτωση που συζητάμε. Μπορεί κάποιοι να έχουν ε, θρησκευτικούς ε, σκοπούς και να νομίζουν ότι υπηρετούν το δίκαιο και διορθώνουν τις αδικίες. Όμως, ε, επειδή υπάρχει και η κρίση στην Ευρώπη, πολλοί από τους νέους αυτούς είναι άνεργοι και απελπισμένοι. Μπορεί αυτό να είναι μια εξήγηση για την πορεία που παίρνουν. Αλλά και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε ότι κάποιοι απειλούν να πάρουν πίσω την υπηκότητα, να θα την ηθαγένεια των ανθρώπων αυτών εφόσον επιστρέψουν. Αυτό μου φαίνεται τελείως ε, βλακώδες. Μου φαίνεται πραγματικά βλακώδες, δεν έχει κανένα νόημα και θα παραμένω στη γραμμή που και εσείς από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα πρέπει να δικαστούν, να δικαστούν ως εγκληματίες, ναι, ως μέλη μιας δημοκρατικής οργάνωσης, ναι, αλλά τώρα να του αφαιρέσει κανείς την ηθαγένεια τι θα πει αυτό. Απλώς θα μετατοπίσουμε το πρόβλημα στην γειτονιά μας. Και δεν θα φύγει καν την επικράτεια της Ευρώπης φαντάζομαι. Το άλλο ερώτημα που θέλω να σας ρωτήσω. Και επειδή κάνατε κάποιες συγκεκριμένες διευκρινήσεις, φαντάζεστε ότι τα Γκουαντάναμο θα πολλαπλασιαστούν. Όλη αυτή η σύγχυση που είναι τελείως παράνομη και την οποία διοργάνωσαν κάποιοι από τους ε, συνεργάτες μας ε, για τον οποίο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να ενισχύουμε ενδεχομένω περισσότερο από κάποιες άλλες περιπτώσεις και το κράτος δικαίου στην περίπτωσή τους. Την διοργάνωσαν λοιπόν και την άφησαν να πολλαπλασιαστεί. Επιβεβαίωνετε ότι γι' αυτό το τονίσατε. Και επίσης τι μπορείτε να κάνετε για να βεβαιωθούμε ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι μυστικές μας υπηρεσίες και η διάρθρωση της συνεργασίας τους μεταξύ τους ε, να βελτιωθεί, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και εδώ έχουμε πολλά προβλήματα, Ιδίω εν ώψη των, ε, υπό το των απειλών που αντιμετωπίζουμε τώρα. Χρειάζεται πολύ πιο απτή συνεργασία στο επίπεδο των ε, μυστικών υπηρεσιών και με δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία και βάσει βεβαίως των κανόνων που ισχύουν. Όπως προκύπτει και από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Γκόμες, ο κύριος Τάνοκ. Σας ευχαριστώ. Δεν ε, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά όσο και να σέβομαι την Άννα και παίρνω στο σοβαρά την αποψή της, δεν μπορώ να αποδεχτώ το ότι περιγράφουμε ως ε, ε ηλίθιο τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Ντέβιτ Κάμερον υπερασπίζει την ε, αρχή της στέρησης ε, της ηθαγένειας από τους υπηκόους που, του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν βγει στο εξωτερικό και έχουν διαπράξει εγκλήματα στο όνομα της ίσης. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και ποινική δίωξη. Δεν δέχομαι ότι η ενεργεία αποτελεί αιτία τρομοκρατίας, Άννα. Θα ήθελα να θέσω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Στο ένα μπορεί να μην μπορείτε να απαντήσετε. Στη Βρετανία έγινε προσφάτω μία συζήτηση και μία ψήφο στο House of Commons σε ό,τι αφορά το δικαίωμα να γίνονται ε, ε, επιθέσεις κατά της του ISIS. Extended from Iraq, where clearly Britain... Οι επιθέσεις αυτές από το Ιράκ, από, το, από ε, στη Συρία και από άλλε χώρες χωρίς την ε, έγκριση του κυρίου Ασάντ παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις προέρχονται από την Συρία και άρα μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι το Ιράκ ε, ήταν σε άμυνα σύμφωνα με το χάρτη της Ευρωπαϊκής του, του ΟΗΕ αλλά επίσης αναφέρεται το δικαίωμα προστασίας των πολιτών του από φρικαλαιότητες ε, και οποιοδήποτε έχει δικαίωμα και μέσω να το πράξει αυτό έχει δικαίωμα να παρέμβει. Αυτό νομίζω ότι σημαίνει ότι μπορεί όντως να μην χρειαζόταν η έγκριση του κυρίου Ασάντ. Έχετε μία άποψη ή δεν σα απασχολεί αυτό. Κάτι άλλο. Αναφερθήκατε σε ημάμιδες που έρχονται από την υποσαχάρια Αφρική. Καλωσορίζω αυτή, το, αυτή την κίνηση. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Κάποιες χώρες, το Κατάρ για παράδειγμα, που έχουν σαλαφιστική ιδεολογία, κάνουν πως δεν βλέπουν ή υποστηρίζουν άμεσα τρομοκρατικές οργανώσεις. Τι μέτρα λοιπόν μπορεί να λάβει ο ΙΕ για να ασκήσει κριτική στα κρατημέλη του αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και να τα αποθαρρύνει από τέτοιες πρακτικές. Ευχαριστώ κύριε Μωράες, αν θα θέλετε να πάρετε την Προεδρία και να δώσετε το λόγο. Έχουμε άλλα 15 λεπτά, 20 μάξιμου λόγω των διερμηνέων. Ναι. Μου φαίνεται τα δύσκολα, λέει ο κύριο Μωράες. Είναι πολύ περίεργο και το σύστημα ρύθμισης ε, της ΑΦΕΤ. Μάλιστα. Κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, ε, δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί η ΑΦΕΤ, αλλά εμείς θέτουμε μόνο μία ερώτηση. κάνω πλάκα, Charles. Βρετανικό φλέγμα. Ερωτώ λοιπόν, δεν είναι πολιτικό το ερώτημα, είναι πρακτικό το ερώτημα. Από πλευρά σου, πείτε μας. Τι πιστεύετε για την οδηγία διατήρησης δεδομένων και την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τι είπατε, α, μάλιστα, για την διατήρηση δεδομένων. Δεν κάνω πολιτικό σχόλιο. Ένα κρατός μέλος τουλάχιστον. Αναγκάστηκε να προσαρμόσει την νομοθεσία του για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατική απειλή. Είναι αυτό κάτι γενικότερο. Εμείς στο Κοινοβούλιο είχαμε την αίσθηση ότι δεν υπήρχε ανάγκη να συλλεχθούν τόσα προσωπικά δεδομένα για να αντιμετωπιστεί η απειλή της τρομοκρατίας. Ποια είναι η προοπτική που έχετε λοιπόν εκτός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για τέτοια αναγκαιότητα. Ή πιστεύετε ότι ήταν σωστή αυτή η απόφαση. Θα ήθελα να ακούσω την απόψή σας και Στη συνέχεια να δώσω το λόγο στον κύριο Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Λαμπόρτ που είστε εδώ. Είναι μεγάλη μας τιμή να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, με μια ε, κοινή ε, συνεδρίαση και των δύο επιτροπών που ασχολούνται με την εξωτερική διάσταση της ε, καταπολέμηση με την οποία ασχολείται η ΑΦΕΤ, και την εσωτερική, που είναι ευθύνη τη ε, ΛΥΜΠΕ. Η Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων Δικαιοσύνη και δικαιωμάτων των πολιτών ε, απορρίπτει την ε, να δράσει κατά, λες και πρόκειται για νομοθέτη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια νομική απάντηση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, και η πρώτη μου ερώτηση προς εσάς είναι ω υπεύθυνο και διευθυντή για την υπηρεσία του ΟΗΕ της καταπολέμηση της τρομοκρατίας και βάσει της πείρα σα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για να ορίσουμε την τρομοκρατία είναι ακόμη πρόβλημα αυτό. Ε, βέβαια όλοι έχουμε καταλάβει πλέον ότι η τρομοκρατία έχει να κάνει με τους, όχι μόνο με τους ε, σκοπούς που κανεί ε, ευαγγελίζεται αλλά κυρίω με τα μέσα που χρησιμοποιεί, δηλαδή τις αδιάκριτες δολοφονίες, τις επιθέσεις. Οι στόχοι όμως, ε, είτε είναι ιδεολογικοί είτε η θρησκευτική παστικοποίηση ακόμη μετράνε. Είναι λοιπόν ένα συνδυασμό που είναι φρικτός και μας απειλεί ήδη στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα, στα σύνορα ε, Τη πρώην Σοβιετική Ένωσης, της ε, Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ε, ο θανάσιμο συνδυασμό εξτρεμιστικών κινημάτων και θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση Με, σε εδάφη της πρώην μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης. Εδώ λοιπόν κάποια μαθήματα μπορούμε να αντιλήσουμε από το παρελθόν. Ποια είναι αυτά τα μαθήματα και πώς μπορούμε να ορίσουμε από νομική σκοπιά στην τρομοκρατία Μία ερώτηση. Είπαμε να ρωτήσουμε μία ερώτηση και τώρα μου δίνεται κακή εικόνα. Εντάξει, μία, αλλά θα είμαι πολύ σύντομο. Είναι ιδιαίτερη ευκαιρία. Λοιπόν, ε, η δεύτερη ερώτηση με αφορά την χρηματοδότηση. Για το Ισλαμικό κράτος δεν είναι πρώτα απ' όλα σφάλμα να το καλούμε κράτος και μετά να έχει χρηματοδοτηθεί από κράτη της διεθνούς κοινότητας. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε, για να, καθορίσουμε, να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση του ISIS και τις τρομοκρατικές του ενέργειες. Και τρίτη ερώτηση. Χρησιμεύει σε τίποτα το PNR. Έχει αποδώσει κάτι. Μας βοηθάει σε τίποτα για να προλάβουμε την τρομοκρατία. Μόλις έκανα μια μεγάλη ομιλία για τη μία ερώτηση μέλος της Λίμπε και εσύ τελικά με διέψευσε πλήρως. Ε, Αλλιώς ο Τσάρλς θα είχε θέσει τέσσερις. Κυρία Λέζινγκ, θα μας βοηθήσετε, ε, αν και είστε άφετο, οπότε μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Και θα ήθελα λοιπόν να, ε, να συμφωνήσω με την ερώτηση του συναδέλφου από τη Λίμπε. Χωρίς τη μαζική υποστήριξη διάφορων κρατών, το ίσις δεν θα μπορούσε να είναι τόσο ισχυρό και τόσο μεγάλο, να αποτελεί τόσο μεγάλη απειλή όσο αποτελεί σήμερα. Θελώδης λοιπόν είναι πάντα οι ενδείξει από διάφορα κράτη αναφέρεται ότι υποστηρίζετε. Ερωτώ λοιπόν εσάς, έχετε πιο ακριβή στοιχεία, ποια κράτη και πώς, με ποιο τρόπο υποστηρίζουν το ίσις. και στη συνέχεια πώς ε, σκοπεύετε, πώς ε, προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την υποστήριξη ε, με εκπροσώπους ενός κράτους που υποστηρίζει ανοιχτά σχεδόν το ίσις. Μιλήσαμε πριν από μισή ώρα με την Τουρκία και αύριο θα γίνει μια ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πρέπει να πω ότι αυτά που άκουσα πριν από μία ώρα με σόχαραν ιδιαίτερος. Δεν νομίζω ότι έφταιγε το γεγονό ότι δεν είχε ώρα στη διάθεσή του ο εκπρόσωπος της Τουρκίας. Σκοπίμως και θελημένα της απέφυγε να μας μιλήσει για το πώς υποστηρίζει η Τουρκία οικονομικά το ίσις και πώς ε, παρέχει και ε, διοικητική αρρωγή δεν ε, αναφέρθηκε καθόλου στο πώς η Τουρκία προτίθεται να αλλάξει την πολιτική της ως προς το θέμα αυτό. Συγκεκριμένο ερώτημα προς εσάς. Συμφωνείτε λοιπόν με την άποψη ότι δεν φτάνει να μείνουμε στα ευγενή και φιλικά λόγια της διπλωματίας και ότι προς τα κράτη αυτά, τα κράτη για τα οποία ξέρουμε, όπως η Τουρκία για παράδειγμα, εσείς ε, ίσως να έχετε και πιο πολλές πληροφορίες, θα πρέπει να ασκήσουμε μεγάλη πίεση. Να συμφωνήσω και με την ερώτηση του κ. Τάνοκ. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις ε, εναέριες επιθέσεις στο Συριακό έδαφος στην επικράτη της Συρίας. Μας καλύπτει η εντολή του ΟΗΕ ή πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ κυρία, την κυρία Λούζικ και τώρα ο κύριος Σεπαϊέν. Η κυρία Σεπαϊέν. Ναι, ναι, ναι. Μην βγάζετε τα ακουσικά σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας ε, για την πολύ λεπτομερή παρουσίαση αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στην αρχή μιλήσατε για την αρχή της μη διάκρισης, ε, αλλά οι εθνικές ε, καταστάσεις ε, κατεπίγουσας ανάγκης είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί να κάνουμε εξαιρέσεις. Τι υπάγεται λοιπόν στο πλαίσιο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση μαζικής παρακολούθησης, όπου γίνεται profiling ε, λόγω του ονόματος, ε, του χρώματος, του δέρματος του καθενός, του τραπεζικού του λογαριασμού. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί στο παρελθόν και δεν θέλουμε να ξαναδούμε να συμβαίνουν. Και όπω είπα, όπως είπε και η Άννα Γκόμες προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν να χάσει κανείς την υπηκότητά του, ακόμα και την δεύτερη υπηκότητά του. Όταν ε, μιλάμε για τους μαχητές που αναφέρθηκαν και αυτό ενδεχομένως να θεωρήσει και να οθήσει τις χώρες να χαρακτηρίσουν το φαινόμενο αυτό ως κατάσταση εκτάκτης ανάγκης. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πόσοι είναι και όταν επιστρέψουν είναι ένοχοι εγκλημάτων είναι κατηγορούμενοι τέτοιων εγκλημάτων. Θα πρέπει να υπάρξει έρευνα για τα εγκλήματα αυτά. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε απλά ότι επειδή κάποιος έχει πάει κάπου είναι αυτομάτως ένοχος. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε συναδελφή χρόνο. Αν ε, συμφωνείτε να μην ε, θέλετε πολλές ερωτήσεις γιατί είναι μεγάλος ο κατάλογος ακόμα. Επόμενος ομιλητής η κυρία Γουινμπέρκ του EFTD και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Μπόρτ, που ήρθατε εδώ. Απαντήσατε σε κάποιες από τις ερωτήσεις μου, ούτως ή άλλως, αλλά ήθελα λίγες περισσότερες λεπτομέρειες το πλαίσιο στο οποίο βλέπουμε πλέον να περιέρχονται η Συρία και το Ιράκ. Έχουμε κάποια θέματα αρμοδιοτήτων όπως βλέπουμε εδώ. Εάν όμως δεν κάνουμε κάτι και από νομική σκοπιά, αν δεν λάβουμε κάποια μέτρα, δεν θα εμποδίσουμε να πηγαίνουν προ τα εκεί και οι ξένοι μαχητέ λόγου χάρη. Είδαμε τώρα το ψήφισμα του 29, το ψήφισμα 2178 και τον αντίστοιχο τρόπο καταπολέμησης τη δημοκρατίας των ΗΠΑ στο άρθρο 2 λέει ότι είναι υποχρέωση η καταπολέμηση των τρομοκρατών ακόμη και με συνοριακού ελέγχου ή ελέγχου διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων inter alia, όπω αναφέρει το κείμενο. Πώ μπορείτε αυτό να βεβαιωθείτε ότι θα ισχύσει και στην περίπτωση των τρομοκρατών στο άρθρο 8 του ψηφίσματο, Δεν λέγεται πώ τα κράτη-μέλη θα εμποδίσουν τους δικούς τους τους υπηκόους να, πάνε, να φύγουν από τις χώρες τους για να πάνε να ε, συνεργαστούν με τους τρομοκράτες. Επίσης το ψήφισμα στο άρθρο 4 το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί τα κράτη-μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουν την ρίζοσπαστικοποίηση ή τη στρατολόγηση ή τη χρηματοδότηση από πρώην ε, στρατεμένους. Επίσης, το ψήφισμα του ΟΙΕ ορίζει ότι όσοι συμμετέχουν, χρηματοδοτούν ή ασχολούνται με την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών θα, δικάζονται στα δικαστήρια και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν ποινές καταστολής. Πώς περιμένετε τα κράτη-μέλη ότι θα εφαρμόζουν αυτέ τι ποινές, ε, ε, συνάδελφοι, παρακαλώ, ε, συμπιέστε λίγο τι παρεμβάσεις σα. Πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι. Χρειάζεται μισή ώρα για να απαντήσω σε όλα αυτά. Εγώ είπα στους συναδέλφους να μην ρωτούν ε, πολλαπλές ερωτήσεις, αλλά ο Βρετανός συνάδελφος άλλαξε την ε, ρότα της συζήτησης. Μη με κατηγορείτε, έκανα ό,τι μπορούσα. Εγώ έδωσα καλό παράδειγμα. Είμαι Βρετανός. Έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά ο Βρετανός συνάδελφος με κρέμασε. Η ε, κυρία Σεράια θα ερωτήσει μία ερώτηση, γιατί είναι μέλος της ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά όσα λέτε και νομίζω ότι το γεγονό ότι κάποιε θεμελιώδει αξίε θα τι σεβαστούμε ό,τι και να γίνει είναι κάπω καθησυχαστικό. Ε, ορίζονται και από την ε, χάρτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ΙΕ. Όμω βλέπουμε ένα τεράστιο πρόβλημα δημοκρατία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι από τη μια έχουμε εξτρεμιστικέ δυνάμει εντό αλλά και εκτό των συνόρων μα. Λόγου χάρη ακροδεξιέ δυνάμει οι συζητήσεις λοιπόν στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Εδώ έχουμε δύο παράλληλες κινήσεις, ε, εκτεμιστικές δυνάμεις ε, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά τι θα γίνει αν συνεργαστούν μεταξύ τους. Είναι λοιπόν μια ιδέα αυτό που λέτε, ότι πρέπει τους ε, τους ημάμιδε, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να του αξιοποιήσουμε και για ε, τον αντίστροφο σκοπό, για την διατήρηση δηλαδή τη ορθολογιστική κοινωνία των πολιτών. Από το 2001 ε, οι εξτρεμιστικέ δυνάμει φαίνεται να έχουν ξυπνήσει. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε η κυρία Κιένγκε. Σεσίλ. Ευχαριστώ. Αρχικά δεν θα ζητούσα το λόγο, αλλά πραγματικά ε, εντυπωσιάστηκα και από μία ερώτηση για την αφαίρεση της ε, ειδικότητας. Θα σταθώ σε αυτό το σημείο και μόνο. Ε, ήθελα να μου πείτε τι γνώμη έχετε για την πρόταση αυτή, την αφαίρεση της ειδικότητας σε άτομα που είναι ξένης προέλευσης. Κάποιοι έχουν γεννηθεί στο έδαφος μας και έχουν μεγαλώσει εδώ. Θα τους αφαιρεθεί η υπηκότητα. Πού θα πάνε. Ε, εάν ο νόμος του θεωρεί όλους ισότιμους, το θέμα της αφαίρεσης της υπηκότητας ε, έχει να κάνει μόνο με την ε, προέλευση, προέλευση από την αλλοδαπή. Ιδάλω, είτε είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στον νόμο, είτε υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Ήθελα λοιπόν τη γνώμη σα για τι χώρε που ξαναζούν την ανομία ε, για την ε, ε, υπηκότητα. Θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί ω ένα όπλο ήπιο. Σα ευχαριστώ, Σεσίλ, και τέλο με την αδειά σα να κλείσω, να προσθέσω μάλλον στη λίστα τον κύριο Τιγκράφ, ο οποίος είναι από την ομάδα των Εκτός μικροφώνου, ωστόσο. Er Τρία πράγματα. Οι μεγάλοι πολιτικοί λένε ότι το Ισλαμικό κράτος δεν έχει να κάνει τίποτα με το Ισλάμ. Ο Ομπάμα, ο Κάμερον και εκ παραλλήλου βλέπουμε μεταξύ άλλων ότι στην Ολλανδία οι μυστικές υπηρεσίες λένε ότι τα κίνητα των τζιχαντιστών που πηγαίνουν σε Ισλαμικό κράτος είναι και εξηγούνται μόνο για λόγους ιδεολογίες που είναι βασισμένοι στο Ισλάμ. Και το τρίτο θέμα που βλέπουμε είναι ριζοσπαστικές παστικοί οι μάμιδες στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από χώρες όπως το Κατάρ. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποια είναι η απόψή σας. Πιστεύετε ότι το Ισλαμικό κράτος έχει να κάνει τίποτα με το Ισλάμ ή και μπορούμε στην Ευρώπη μάλλον να κάνουμε τίποτα για την ριζοσπαστικοποίηση αυτή. Μεταξύ άλλων να απαγορεύσουμε να μιλούν οι μάμιδες. Thank you very much, Ευχαριστώ και να δείξω κάποια ζητήματα, λέει ο Πρόεδρος, τα οποία να πω στου συναδέλφους που έχουν μείνει την Πέμπτη ότι είναι σημαντικά τα θέματα αυτά και θέλατε όλοι ασφαλώς να κάνετε σχόλια. Λυπάμαι που σας ε, περικόψαμε το χρόνο ομιλίας. Αν θα θέλετε να απαντήσετε σύντομα. Ξέρω φυσικά ότι είναι αδύνατο αυτό το έργο, αλλά ίσως αν οι συνάδελφοι δεν ε, θεωρήσουν ότι έχει απαντηθεί τα ζητήματα που τους έθεσαν, να απαστείλουν κατηδίαν γραπτά ένα... Να σας επικοινωνήσουν γραπτά με εσάς, αν είναι αυτό μια δυνατότητα, αν το δέχεστε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω για να θέσουμε το θέμα της υπηκότητας. Αν ξαναδιαβάσετε την παράγραφο 8 του ψηφίσματος, τι λέει ότι υπό τον όρο ότι τίποτα δεν θα υποχρεώσει μία χώρα να απαγορεύσει την αποχώρηση ε, από την επικράτειά του επικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν για το θέμα αυτό. Και ξέρετε ότι κατά πάσα πιθανότητα ανάλογα με την απειλή και ανάλογα αυτό σχετίζεται με τα έκτακτα μέτρα και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που ακούσαμε για τη Διεθνή Συνέδρια για τα πολιτικά δικαιώματα και τι πολιτικέ ελευθερίε. Έκτακτα μέτρα μπορεί να ληφθούν, αλλά μόνο σε περίοδου έκτακτη ανάγκη, το οποίο, για να απαντήσω, απειλούν τη ζωή του έθνου βάσει μια επίσημη διακήρυξη. Έκτακτα μέτρα υπόκεινται σε αυστηρού όρου, μεταξύ άλλων ε, στην διατήρηση ορισμένων δικαιωμάτων ανεξαίρετα. Δεν αποφασίζουμε εμείς, λοιπόν, κατά πόσον θα αφαιρεθεί ή όχι η υπηκότητα. Αυτό είναι τόσο εθνική απόφαση. Το Συμβούλιο δεν έχει λάβει δράση. Αντιθέτως, ούτε θέση. Δεν πρόκειται να υποχρεώσει κανένα κράτος. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι παραπάνω από αυτό αναφορικά με τον ορισμό του της τρομοκρατίας. Για μας τα Ηνωμένα Έθνη τα πράγματα είναι απλά. Φυσικά, ο ορισμός της τρομοκρατικής ενέργειας είναι μια ενέργεια η οποία ορίζεται στα 18 μέσα, τα οποία έχει εγκρίνει ο ΙΕ. Και θα επανέλθω στα πρώτα μου καθήκοντα ως δικαστής του ακριτικού δικαστηρίου ε, για ποινικά ζητήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικός ορισμός του, της τρομοκρατίας. Μην κάνετε τέτοια απόπειρα. Αυτό το ζητώ πάντα. Γιατί, γιατί εδώ μιλώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και θα ήθελα να πω το εξή. Αν υπάρχει γενικό ορισμό τη τρομοκρατία, αυτό τι σημαίνει ότι κινούμαστε κατά τη αρχή τη νομιμότητα. Είμαστε κατά τη αρχή τη νομιμότητα ορίζονται οι πράξεις της τρομοκρατίας και μετά από χρηματοδοτικής άποψης μπορεί να υπάρχουν οργανώσεις που να υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες, αλλά να συσχετίζονται με ενέργειες αυτό. Φυσικά υπάρχει ορισμός για το τι αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι διαφορετικό. Υπάρχει σχετικός κατάλογος. Και εδώ θέλω να απαντήσω σε αυτά που ακούσαμε για την υποστήριξη του ίσης. Είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει τη δομή ενός κράτους, όπως είπα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί κράτος γιατί η δάλος ε, είναι τελείως λανθασμένα τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει συγκαταλέξει το ίσης στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Το γεγονός αυτό από μόνο του αρκεί για να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Και αυτό ασφαλώς συνδέεται με το γεγονός ότι τα στρατιωτικά μέσα που έχουν ληφθεί κατά του ίσης. Είπατε ότι υπάρχει ανάγκη ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Στέφαν Ταμιστούρα για το κομπάνι, τι είπε, χρειάζεται να υπάρξει άλλη μια στρεμπρένιτσα. Αυτό είπε, αυτό είπε, σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό ήθελα να παραθέσω. Και τέλος, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα. Χρηματοδότηση του ίσης και όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων. Καταρχάς υπάρχει ένα κίνημα και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ένα κίνημα κάποιων κρατών μελών και μερικά από αυτά που αναφέρατε για να εναρμονιστούν με τη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι σαφές ότι όλα τα κράτη τα οποία εκπροσωπούνται από τους ηγέτες τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας κινούνται προς την ίδια γραμμή γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η απειλή είναι απειλή για όλους, ούτε καν μια απειλή μόνο για την Ευρώπη, για τα Ηνωμένα Είναι απειλή για όλους. Και τέλος. Υποδείξατε κάτι πολύ σωστό, Πρόεδρε. Είπατε ότι δεν πρέπει να αντιδράμε, πρέπει να δράμε. Τα μέτρα χρηματοδότησης τώρα. Κανείς δεν ανέφερε την παράγραφο αυτή, δεν την παρέθεση, αλλά υπάρχει και η παράγραφος 6 του ψηφίσματος, η οποία τι λέει ότι όσοι χρηματοδοτούν τους μαχητές αυτούς θα υποστούν μέτρα και είμαι βέβαιος το FTF ε, θεωρώ είμαι και με βέβαιος ότι θα πάρει τα σχετικά μέτρα. Και όπως είδαμε και στο παρελθόν για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αυτό θα πάρει χρόνο τα μέτρα αυτά. Δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι τα κράτη και η διεθνή κοινότητα μπορεί να πάρει τα μέτρα αυτά γρήγορα και άμεσα για την διατήρηση τώρα των προσωπικών δεδομένων, το PNR. Να πω ένα πράγμα. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πιο δεσμευτικό και περιοριστικό αν υπάρξει ευρωπαϊκό σύστημα γιατί εσείς ασχολείστε πιο πολύ με το θέμα των ελευθεριών των κρατών μελών. Αυτά με ρωτήσατε, αυτό ήθελα να σας απαντήσω. Τα δεδομένα είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο. Οι μυστικές υπηρεσίες δεν αποτελούν πρόβλημα Είμαι σίγουρο ότι συνεργάζονται άριστα. Το θέμα είναι να προσαχθούν σε δίκη αυτοί οι άνθρωποι και προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει κάτι το βάσιμο προκειμένου να μπορέσουμε να τους σταματήσουμε στα σύνορα και να τους προσάγουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό ήθελα να, να τονίσω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σε σχέση με την Επιτροπή μας που εξετάζει και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης, ε, όλα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που προσπαθήσατε να πετύχετε το αδύνατο και να ευχαριστήσω και τους βουλευτές για την υπομονή του σήμερα. Κύριε Πλένκοβιτς, θέλετε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι, για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον προσκεκλημένο μας. Πέρα στη συνεδρία σας. Ευχαριστώ κύριε Μωράη, ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 3 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ.